the European Centre for the Development of Vocational Training, and the Secretariat has drawn up a feedback note that you can read in today's meetings documents. Approval of meetings of minutes. Έκριση, μάλλον δεν ακούγεται το μικρόφωνο. Έγκριση των πρακτικών της 25ης Ιανουαρίου, 17-18 Φεβρουαρίου, και 23 Φεβρουαρίου του 2016. Μπορούμε να τα εγκρίνουμε. Και έτσι φτάνω στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Και καλωσορίζω θερμά τους επιτρόπους κυρία Τάισεν και κύριο Ναύρατζες. Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ. και προσβλέπουμε σε μια πολύ καλή ενημερωτική, εμπλουτιστική και εμπνευστική συζήτηση. Και του των λεχθέντων δίνω τον λόγο στη συνάδελφο κυρία Κώστα για να κάνει την εισαγωγή. Έχετε τον λόγο παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, abbiamo Πενσίδη αγαπητοί συνάδελφοι, σκεφτήκαμε όλοι σαν Επιτροπή Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Εργασίας και με την παρουσία των δύο Επιτρόπων εδώ, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση αναφερόμενας σε πρόσωπα τα οποία νομίζω μας ε, αφορούν όλους ε, τους 13 υποτρόφους Εράσμους που βρήκαν το θάνατο στην Ισπανία πριν από λίγες εβδομάδες. Φυσικά τιμήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και τους νεκρούς των Βρυξελών και σήμερα μαθαίνουμε ότι υπάρχουν πάλι πάρα πολλοί νεκροί στη Μεσόγειο μετά από ναυάγια. Έβας αναφερόμαστε εδώ στα 13 κορίτσια μάλιστα από εντελώς διαφορετικές εθνότητες ε, ζούσαν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία στην Καταλωνία και νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα, ευρωπαϊκού τύπου πένθος. Ελπίζουμε να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να δίδονται περισσότερο εγγυήσει ασφαλείας στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του Εράσμους και το Εράσμος πρέπει να είναι κάτι το θετικό, μια θετική εμπειρία, μια εμπειρία χαράς και στο όνομά τους θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες γύρω από το Εράσμος. Και γι' αυτό να σας ζητήσω παρακαλώ ενός λεπτού συγγύη προς τιμήν των νεκρών κοριτσιών την Βαλεντίνα, την Έλενα, την Ελίζα, την Λουκριτία, τη Σερένα, την Φραντσέσκα, την Ελίζα, την Μοκίνα, την Κλοέ, την Βερόνικα, την Φόναμαντ, την Τζούλια και την Κριστίνα. Και πάλι λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την πρωτοβουλία να κάνουμε την ακρόαση για το θεματολόγιο για τις δεξιότητες αφορά την Επιτροπή Απασχόλησης και την Επιτροπή Πολιτισμού. Δεν χρειάζεται να το πούμε βέβαια εδώ, αλλά θα το επαναλάβω όπως και να έχει. Πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες για το μέλλον της αγοράς εργασίας, οι δεξιότητες, τα προσόντα έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τις εργασίες μας και ιδιαίτερα θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την πρωτοβουλία αυτή ώστε να εξασφαλιστεί η μόρφωση και οι δεξιότητες για όλους. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν ακόμη Είναι απαράδεκτο στην εποχή μας να γεννιέται κάποιος και να μην μάθει ποτέ ούτε να μετράει ούτε τα να διαβάζει σωστά. Αυτό συμβαίνει ακόμη και σε περιοχές της Ευρώπης και αποτελεί όνειδος. Από αυτό ξεκινούμε. Αυτή είναι η εφετηρία μας, αλλά προχωρούμε περισσότερο ακόμη. Και αρχίζοντας δίνω το λόγο στην κυρία Τάισεν για μια παρουσίαση αυτού του κέριου για τις επιτροπές μας θέματος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Ευρωβουλευτές. Χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι εδώ στο σώμα και πάλι μάλιστα σε μια κοινή συνεδρίαση για τις δεξιότητες. δεξιότητες ήταν το θέμα μια από τις πρώτες μου ε, ομιλίες στην Επιτροπή Πολιτισμού όταν ξαναγύρισα στο Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο του 2015 ως Επίτροπος πλέον και βλέπω ότι έχει ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα για τις εργασίες των Επιτροπών σας. Ιδιαίτερα καλώς ορίζω την έγκριση του ψηφίσματος για τις δεξιότητες της κυρίας Πλούρατς και, της κυρίας, και την έκθεση της κυρίας ε, Νεπαρόριτς για τις ε, δεξιότητες επίσης. Υπάρχουν ε, εκθέσεις που έχουν να κάνουν με το Erasmus Plus για τον περιορισμό των ελλείψεων σε δεξιώσεις, δεξιότητες, αναγνώριση δεξιοτήτων, κατάρτιση προσαρμογή στο πλαίσιο 2020 εν ώψη του νέου θεματολογίου για τις δεξιότητες. Δεδομένου του χρόνου που έχω στη θέση μου σήμερα, θα ήθελα να σας εκθέσω την πρόοδο των εργασιών, των συνομιλιών και να δώσω τις κύριες γραμμές των ιδεών μας για τα πιο σημαντικά θέματα που αφορούν την Ευρώπη, δηλαδή πώς το εργατικό μας δυναμικό θα εξασφαλίσει τις δεξιότητες που χρειάζονται για να παρακολουθήσει την ταχύτητα μεταλλασσόμενη αγορά εργασίας. Ένα νέο θεματολόγιο λοιπόν δεξιοτήτων για την Ευρώπη. Δεξιότητες για την απασχολησιμότητα. Η οικονομική επιτυχία της Ευρώπης σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις δεξιότητες των πολιτών μας. Η μελλοντική μας ανταγωνιστικότητα και η μελλοντική ανάπτυξη εξαρτώνται από τις δεξιότητες ρυθμοί εξελίξεων ε, στην αγορά εργασίας καθιστούν μεγαλύτερη ακόμη την πρόκληση. Η ψηφιακή επανάσταση αναδιαμορφώνει τις θέσεις εργασίας ακόμη. Και ξεκινώντας θέλω να πω ότι δεν βλέπω αντιπαράθεση ανάμεσα στην ιδέα των δεξιοτήτων για τον επαγγελματικό και για τον προσωπικό βίο. Η εξασφάλιση λοιπόν των δεξιοτήτων για όλους είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Ο αναλφαβητισμός, η ανικανότητα σε μαθηματικούς ή άλλους όρους δεξιότητας ε, σημαίνουν και αποκλεισμό, όχι μόνο από την αγορά εργασίας, αλλά και από την κοινωνία και υψηλό κίνδυνο φτώχειας. Θέλω λοιπόν να εξασφαλίσουμε πως όλοι θα έχουν τη δυνατότητα με τις δεξιότητές τους να βελτιώνουν την, ε, τις ευκαιρίες τους για τη ζωή και την απασχολησιμότητα για τις θέσεις εργασίας λοιπόν, για την δυνατότητα μετάβασης από τη μία θέση εργασίας στην άλλη, επικοινωνία και προσαρμογή σε νέες δεξιότητες. Και πρέπει να καλύψουμε το κενό ανάμεσα στις δεξιότητες των φτωχών και στις δεξιότητες των πλουσίων. Αυτό σημαίνει στενή συνεργασία μεταξύ διαφόρων τομέων της πολιτικής και κυρίως μεταξύ της απασχόλησης και της εκπαίδευσης. Μαζί με τον συνάδελφο Τίμπορ κάναμε συζήτηση με τους υπουργού ε, Παιδείας το Φεβρουάριο στο Συμβούλιο και ο Τίμπορ πάλι ήρθε στο Συμβούλιο των Κοινωνικών ε, Θεμάτων και της Απασχόλησης σε μια συζήτηση πάλι ε, στη δική μας πλευρά. Συνεργαζόμαστε εντατικά με τους συναδέλφους από όλη την Επιτροπή, από όλους τους τομείς εργασίας, για να ετοιμάσουμε μια νέα πρόταση για το θεματολόγιο για τις νέες δεξιότητες. Είναι λοιπόν πολύ ευπρόσδεκτη αυτή η ευκαιρία, κυρίες ε, συμπρόεδροι, να συστήσουμε σήμερα, γιατί πιστεύω ότι μόνο αν συνεργαστούμε στενά στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στις πολιτικές και την αγορά εργασίας θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε και να εξασφαλίσουμε τις μεταρρυθμίσεις εκείνες που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, να εξασφαλίσουμε ευκαιρίες και ισονομία, ισότιμη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Είναι λοιπόν ε, μεγάλες προκλήσεις. Ένα στους πέντε Ευρωπαίους, 70 δηλαδή εκατομμύρια Ευρωπαίοι, έχουν δυσκολία να διαβάσουν, να γράψουν, αλλά και να κάνουν απλούς υπολογισμούς ή να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικά μέσα. Και όμως τα ηλεκτρονικά μέσα είναι απαραίτητα για τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ε, αναγκάζονται να δεχθούν θέσεις εργασίας χωρίς να έχουν ε, που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους ε, δεξιότητες. Ένα 30% είναι σε θέσεις εργασίας που δεν χρειάζεται ε, πανεπιστημιακό πτυχίο. 40% είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν 40% των θέσεων εργασία είναι αυτέ που δεν καλύπτονται από επαρκή προσόδα και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν, τη δυνατότητα, δεν έχουν ε, συμφωνία ως προς την αξιολόγηση της θέσης τους. Αλλιώς την βλέπουν εκείνοι και αλλιώς την βλέπει ο εργοδότης. Πολλά λοιπόν μένουν να γίνουν και επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω κάποιους τομείς τους οποίους βρίσκω ότι μπορεί μια, ένα τέτοιο θεματολόγιο για τις δεξιότητες να αποδώσει. Καταρχάς θα πρέπει να βελτιωθούν τα επίπεδα των δεξιοτήτων. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε δηλαδή ότι ο καθένας θα έχει και τη μόρφωση και τις βασικές υπολογιστικέ δυνατότητες και όλες τις δεξιότητες για την αγορά εργασίας και την ε, καθημερινή ζωή. Νέα συστήματα λοιπόν εκπαίδευση και κατάρτιση που θα πρέπει να αξιοποιηθούν, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται και νέε ευκαιρίε για εκείνου οι οποίοι έχουν ήδη προχωρήσει στη ζωή. Χρειάζονται υψηλές δεξιότητες όλο και περισσότερο. Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να τις ε, αποκτούν κατά τη διάρκεια των ε, σταδιοδρομιών τους και η ταχύτητα των αλλαγών σημαίνει ότι πολύ σύντομα δεξιότητε θεωρούνται πεπαλαιωμένε και χρειάζεται να αντικατασταθούν από νέε τεχνολογίε, νέου τρόπου εργασία. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, πρέπει να δώσουμε λύσει ώστε να μπορούν οι πολίτε και να επικαιροποιούν και να αναβαθμίζουν τι δεξιότητέ του σε όλη την επαγγελματική του ζωή. Εξετάζω λοιπόν το δυναμικό για μια εγγύηση δεξιοτήτων που θα έδινε καθοδήγηση προ τα κράτη-μέλη για το πώ μπορούν να ενισχύουν την πρόσβαση και την απόκτηση δεξιοτήτων για τους ενηλίκους εκείνους που δεν έχουν επαρκή, επαρκή κατάρτιση. Και από την εκπαίδευση και από την αγορά εργασίας μπορούμε να βοηθήσουμε στην επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας. Δεύτερον, η ενίσχυση της ποιότητας και της ελκυστικότητας της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευση, ώστε να είναι οι επιλογές των νέων και των γονέων τους οι πρώτες αυτές που θα ακολουθήσουν και όχι κάποιες ε, ιστερότερες. Η ε, εμπλοκή και του επαγγελματικού κόσμου επίσης μπορεί να βοηθήσει, του επιχειρηματικού κόσμου, για να προσδιορίσουμε υψηλού επίπεδου κατάρτιση και βέβαια μαθητεία. Και τρίτον θα πρέπει για να καλυφθούν ε, τα ελλείμματα και οι αναντιστοιχίες στις δεξιότητες να προβλεφθούν και να ε, εντοπιστούν εγκαίρως οι ανάγκες σε δεξιότητες και να εξασφαλιστούν δεξιότητες ορατές για όλους. Ιδιαίτερα με την κρίση, την προσφυγική και τη μεταναστευτική αυτό καθίσταται ορατό και απαραίτητο. Μια καλύτερη κατανόηση των δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για μια απρόσκοπτη ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας και για την ε, είσοδο στις ε, επαγγελματικέ δραστηριότητες του μέλλοντος. Ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στην επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μέσα στην Ευρώπη από ό,τι δείχνει μελέτες, όπου 17% των Πολωνών πτυχίουχων που θέλουν να ανοίξουν δική του θέλουν δική τους επιχείρηση, ενώ μόνο 3% των Αυστριακών, Γερμανών ή Δανών ε, συνομιλίκων τους ε, μπορεί να δείχνουν τέτοια πρόθεση. Πώς λοιπόν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ώστε να μπορεί κανείς να έχει στον τον καλύτερες δεξιότητες για να θεωρεί ότι είναι σε θέση να ξεκινήσει μια νέα ε, και νεοφύη επιχείρηση. Οι επιλογές λοιπόν είναι πολλές και πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε τη δουλειά για, σε όλους τους τομείς πολιτικής για να οδηγηθούμε σε μια πραγματική αλλαγή πολιτικής. Οι αλλαγές λοιπόν στην αγορά εργασίας όταν δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν σε δεξιότητες και εκπαίδευση θα οδηγήσουν απαραίτητα ε, εξάπαντο σε ελλείμματα. Μαζί με τους συναδέλφους ε, είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε πλήρως προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή. Στη διάθεσή μας έχουμε σημαντικούς πόρους, ώστε αυτό το θεματολόγιο να υλοποιηθεί με επιτυχία. Είτε πρόκειται για τα 27 δισεκατομμύρια ευρώ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση και τη διαβίου μάθηση. Είτε πρόκειται για το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Ταμείο ή το πρόγραμμα Erasmus Plus πρόκειται για πόρους που μπορούν να φέρουν σημαντικές αλλαγές στις ζωές των πολιτών. Περιμένω με χαρά να ακούσω τις δικές σας απόψεις και προσβλέπω στη συνεργασία μας σας για να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή τη σχετική με τις δεξιότητες. Είναι καθήκον μας. Το οφείλουμε προς τους νέους, προς τους νέους πτυχιούχους που έχουν μείνει σε μια χαμηλών απαιτήσεων θέση εργασία, ε, εκείνους τους μηχανικούς των οποίων οι δεξιότητες θεωρούνται πεπαλαιωμένες γιατί έχουν προχωρήσει τεχνολογίες προς ε, νέους ή νέες που δεν μπορούν επειδή δεν έχουν επαρκείς ε, γνώσεις και δεν είναι αρκετά κατηρτισμένοι να προχωρήσουν περισσότερο στη ζωή τους. Όλοι μαζί λοιπόν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Τάισον. Να βάζει, να βάζει, το Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βλέπω και τις δύο επιτροπές να συνεργάζονται πάνω σε αυτό το σημαντικό θέμα, όπως ε, κάνω εγώ και η Μαριάν. Η, ε, η ατζέντα αυτή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ανάλογα από τους δικούς μας θεσμούς. Τόσο η εκπαίδευση και η αποσχόληση παίζουν έναν ιδιαίτερο σημαντικό ρόλο εδώ πέρα. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με ένα ερώτημα. Τι είδους εκπαίδευση είναι αυτή που θέλουμε να έχουμε τα επόμενα χρόνια και τι είδους κοινωνία οροματιζόμαστε. Ε, βλέπουμε ένα αυξανόμενο χάσμα μεταξύ ανθρώπων που έχουν υψηλή κατάρτιση και αυτούς που δεν έχουν τα εκπαιδευτικά συστήματα τα οποία επικεντρώνονται σε ένα περιορισμένο δίκτυο ικανοτήτων με αποτέλεσμα να παρέχονται αυτά μόνο σε ένα ορισμένο αριθμό ε, ανθρώπων για προς όφελος συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Για μένα λοιπόν η απάντηση είναι ξεκάθαρη τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη θα πρέπει να έχουν μια διτή αποστολή. Από τη μία πλευρά θα πρέπει να ανταποκρινόμαστε καλύτερα και πιο άμεσα στις ανάγκες τη αγορά εργασία και ταυτόχρονα να παράσχουμε στους νέους ανθρώπους τις ε, αξίες και τις ικανότητες ούτω ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται και να ενσωματώνονται στην κοινωνία. Και για ποιο λόγο όλο αυτό. Διότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να παραμείνουν απασχολήσιμοι ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να συνεισφέρουν. Νωρίτερα φέτος η Μαρία και εγώ είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε ε, το ζήτημα της, ε, του θεματολογίου των δεξιοτήτων με τους Υπουργούς Απασχόλησης η κυριαρχούσα άποψη ήταν ότι οι δύο αυτές πλευρές ήταν πάρα πολύ σημαντικές ε, και ε, συνάδουν. Το θέμα δεν είναι να, ε, να... επιλέξουμε το μεν το δε. Πιστεύω ότι όλοι σας θέλετε ανεξάρτητους πολίτες οι οποίοι έχουν μια εργασία που τους ολοκληρώνει και για να επιτύχουμε αυτό το στόχο θα πρέπει να αυξήσουμε το επίπεδο κατάρτισης και εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη και θα πρέπει να διασφαλίσουμε το ότι νέοι άνθρωποι αναπτύσσουν ένα δίκτυο ε, ικανοτήτων από μικρή ηλικία και χρειαζόμαστε μια δέσμευση για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης που είναι σημαντική για την βελτίωση της κατάρτισης και της εκπαίδευσης. Από πού λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε η ανάπτυξη κατοτήτων θα πρέπει να ξεκινήσει νωρίς, ε, ήδη από το δημοτικό και τη, δευτερο, ε, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά να συνεχίζεται και αργότερα με τη διαβίω εκμάθηση, τόσο ε, μέσω της επίσημης αλλά και της ανεπίσημης εκπαίδευσης. Τι εννοώ συγκεκριμένα. Αποδείξεις δείχνουν ότι μια πρόορη έναρξη οδηγεί σε καλύτερη απόκτηση των εικονιτήτων και αυτό ισχύει ιδιαίτερως για παιδιά τα οποία έρχονται από, ένα, από οικογένειες που δεν είναι τόσο τυχερές θα πρέπει να προωθήσουμε τις βασικές διεξιότητες πέραν της ανάγνωσης και του αριθμητισμού. Όμως οι ψηφιακές ικανότητες είναι επίσης απαραίτητες ικανότητες. Θα πρέπει να παράσχουμε τους όλους με τις αναγκαίες τεχνολογικές δεξιότητες σε μια κοινωνία η οποία είναι όλο και πιο ψηφιακή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ούτω ώστε να αποτρέψουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό. Δεύτερον, θα πρέπει να δώσουμε στους νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια επιχειρηματική εμπειρία κατά τη διάρκεια της, ε, των σχολικών τους χρόνων. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια συγκεκριμένη δράση σε αυτό, ούτως ώστε οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να ε, ασχολούνται τουλάχιστον μία φορά ε, στον τομέα της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε συνεργασίες με επιχειρήσεις ε, και τους ε, εκπαιδευτικούς φορείς. Όλοι οι παράγοντες της αγοράς εργασίας θα πρέπει να συμμετάσχουν ώστε να κλείσουμε το χάσμα ικανοτήτων. Τρίτον, θα πρέπει να υπάρξει ένα μεγαλύτερο εύρος ε, δεξιοτήτων για τη ζωή. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε, να διδάξουμε στους νέους Ευρωπαίους να μπορούν να στέκονται στα δυο τους πόδια, να βελτιώσουν την ικανότητά τους, την, ικανότητά τους, την κριτική τους σκέψη αλλά και την ομαδική συνεργασία. Όλα αυτά αφορούν τόσο τη στάση αλλά και τις ικανότητες Όλα αυτά θα διασφαλίσουν ώστε οι νέοι άνθρωποι να γίνουν υπεύθυνοι, ευέλικτοι, προσαρμόσιμοι και στη συνέχεια να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις ε, καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας τους και της ζωής τους. Σε αυτό το πλαίσιο η διδασκαλία των κοινωνικών και των πολιτικών ικανοτήτων είναι σημαντική τόσο για τους νέους Ευρωπαίους όσο και για τους μετανάστες ώστε να μπορέσουν να ενσωματωθούν στην κοινωνία αλλά και στην αγορά εργασίας. Αυτά είναι χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν την Ένωσή μας. Θα αναθεωρήσουμε λοιπόν το πλαίσιο των βασικών ικανοτήτων, το οποίο υιοθετήθηκε από κοινού πριν από 10 χρόνια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη το οποίο περιλαμβάνει τις ικανότητες και τις δεξιότητες οι οποίες απαινούνται. Η ατζέντα λοιπόν, ε, το θεματολόγιο δεξιοτήτων είναι σημαντικό για να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη, ούτως ώστε να βελτιώσουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ενώ τέλος οι δεξιότητες αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές σε μια ψηφιακή καινοτόμα ε, οικονομία θα πρέπει λοιπόν η, ανώτερη, η ανώτατη εκπαίδευση να, γίνει, ε, να την προσαρμόσουμε καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η μεταρρύθμιση λοιπόν της ανώτητης εκπαίδευσης θα είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του θεματολογίου. Ενώ επίσης ε, θα πρέπει να ελέγχουμε καλύτερα την αποσχολησιμότητα των αποφύτων ώστε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα σχετικά με το πώ χρησιμοποιούν οι απόφοιτοι τι ικανότητε που αποκτήσαν. Το θεματολόγιο θα πρέπει να έχει μια μακροπρόθεσμη στόχευση ούτως ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά ενώ επίση θα πρέπει να αποτρέψουμε τη δημιουργία νέων κενών σε 10 με 15 χρόνια από τώρα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει να ορίσουμε πιο ξεκάθαρα την κατάσταση και να βρούμε ποιε είναι οι ικανότητε, οι οποίε απαιτούνται για μια οικονομία η οποία αλλάζει συνεχώ. Και επίση θα πρέπει να απευθυνθούμε σε όλου του ανθρώπου, ακόμα και αυτού οι οποίοι έχουν χαμηλή εκπαίδευση, ούτω ώστε κανένα να μην μείνει απ' έξω. Το θεματολόγιο δεξιοτήτων είναι ένα μεγάλο έργο. Το πακέτο λοιπόν το οποίο θα παρουσιάσουμε σύντομα θα είναι μονάχα η έναρξη μιας σειράς πρωτοβουλειών που θα εφαρμοστούν κατά τα επόμενα χρόνια. Ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία εμπιστοσύνη με ανθρώπου οι οποίοι δεσμεύονται και ασχολούνται. Άρα, υπομονώ να ακούσω τι απόψει σα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στον πρώτο γύρο ερωτήσεων και θα δώσω το λόγο για 1,5 λεπτό στον ε, ε, συντονιστή του EPP. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους δύο επιτρόπους για την παρουσία τους και την παρουσίασή τους. Η κυρία Τάισεν αναφέρθηκε στο θέμα ακριβώς των ικανοτήτων και της απόκτησης ικανοτήτων. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να καταστήσουμε εύκολο για τους πολίτες να προχωρήσουν και σε μορφές αυτοαπασχόλησης. Ε, το θέμα της αυτοαπασχόλησης είναι ένα επιπλέον, μια επιπλέον δυνατότητα. Πώς μπορούμε όμως εμείς να βοηθήσουμε τους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα απασχόλησης να περάσουν από την ιδιότητα του μισθωτού, του αμοιβωμένου, στην ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που βρίσκεται σε εκκρεμότητα είναι το θέμα των ικανοτήτων και των γνώσεων των ανθρώπων οι οποίοι είναι άνω των 50. Everybody, okay. Ε, ε, thank you. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Φερχάη, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Επιτροπή Απασχόλησης, ε, θα ήθελα Επιτροπή εκπαίδευση. Ε, θα πρέπει νομίζω να μην αποκοπεί ο ένας κλάδος από τον άλλον η απασχόληση από την εκπαίδευση και βλέπουμε ότι υπάρχει αυτός ο συνδυασμός σε πολλά κράτη, υπάρχει η εμπλοκή της ε, βιομηχανίας, του βιομηχανικού κλάδου και των επιχειρήσεων στην ε, σχολική σταδιοδρομία και αυτό θα πρέπει να το προαγάγουμε περισσότερο. Σε κάποια κράτη προχωρεί καλά, σε κάποια άλλη όμως είναι περισσότερο εσωτερική οργάνωση του σχολείου. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, εφόσον όμω η κατάρτιση που προσφέρει το σχολείο είναι προσανατολισμένη προ την αγορά εργασία και επιτρέπει στου νέου να αποκτήσουν τι δεξιότητε που θα χρειαστούν και στη συνέχεια. Ωστόσο, συχνά μέσα στα σχολεία και τα κέντρα κατάρτιση δεν αναπτύσσονται επιχειρηματικέ ε, δραστηριότητε, δεν είναι κατάλληλα καταρτισμένοι καν οι δάσκαλοι για να τα προσφέρουν στου μαθητέ του. Και σε αυτό νομίζω θα πρέπει να αναπτύξουμε σε πολλαπλές ε, διόδους τη δραστηριότητά μας. Η τεχνολογία επίσης μέσα από τις δεξιότητες της ε, πληροφορικής και της τεχνολογίας θα πρέπει να προαχθεί περισσότερο σε ορισμένες χώρες κυρίως, όπου θα χρειαστεί και οι δάσκαλοι να καταρτιστούν, να μάθουν να χρησιμοποιούν τα διάφορα μέσα της τεχνολογίας, το ίντερνετ, και βεβαίως μπορεί σε ορισμένες χώρες αυτό να εκφράζεται ως ε, επιθυμία αλλά δεν αποτελεί πάντα πραγματικό, πραγματικότητα η δυνατότητα αξιοποίηση τεχνολογίας και τη ανάπτυξη των δεξιοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα και στις ε, πτυχές και στην ε, σχολική αεροδρομία, αλλά και στο διαδικό σύστημα της επαγγελματική κατάρτισης χρειάζεται αυτή τη συνεργασία με τον επιχειρηματικό κλάδο. Ευχαριστώ και εγώ θα εκπροσωπήσω την ομάδα των σοσιαλιστών για την απασχόληση και θα θέσω δύο ερωτήσεις, τις οποίες ήδη έχετε αναφέρει βέβαια. Η πρώτη ερώτηση είναι το θέμα της ευθύνης των εργοδοτών. Στα πλαίσια ακριβώς της ε, των προτάσεων για τις επιπλέον ικανότητες θα πρέπει να βρούμε και τρόπους έτσι ώστε η εργοδοσία να μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των γνώσεων των εργαζομένων τους. Η διαβίου κατάρτιση είναι ένας φορέας και κοινή ευθύνη. Συμμετέχουν φυσικά στα πλαίσια της ανάληψης της συγκεκριμένης ευθύνη και τα συνδικάτα αλλά και οι ομάδες των εργοδοτών και εξωτερικοί οργανισμοί. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα πώς μπορεί να αυξηθεί ο ρόλος των εργοδοτών σε αυτό. Και επίσης τίθεται και το θέμα της πρόσβασης σε αυτές τις διαδικασίες. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το θέμα των ικανοτήτων είναι κάτι το οποίο δεν έχει διανεμηθεί με ισότιμο τρόπο ανάλογα με το σε ποια ομάδα ανήκει κανείς, σε επίπεδο φίλου, σε επίπεδο θρησκευτικό κτλ. Οπότε θα πρέπει να δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να πετύχουμε μια καλύτερη κατανομή των ικανοτήτων ε, στους πολίτες της Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. I think we shall come back so that you can try to ask. Θα επανέλθουμε σε αυτά. Shall we take all? Okay, uh, we have a schedule that forces us to go through all the questions and you. Θα πρέπει να ακούσουμε και τις υπόλοιπες ερωτήσεις και μετά θα δώσετε μια συνολική απάντηση. από την Επιτροπή Πολιτισμού. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen... Κυρία Κάμερα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ ε, για τις εισηγήσεις. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι για το γεγονός ότι η ανταγωνιστικότητα και η οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης εξαρτάται από την εξέλιξη των ψηφιακών ε, δεξιοτήτων. Γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι αυτή τη στιγμή όσοι κάνουν ε, χειρονακτικές εργασίες κρατούν και ένα τάμπλετ στο χέρι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόσκληση θα ήθελα λοιπόν να πω ότι η προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται πάρα πολύ μπροστά ε, στο θεματολόγιο ε, και ότι θα πρέπει να υπάρχει μια επέμβαση η οποία θα ξεπερνάει τις γενναίες. Τα παιδιά θα πρέπει από πάρα πολύ νωρίς να μαθαίνουν τις ψηφιακές δεξιότητες. Ε, αυτό όμως δεν επαρκεί να τους δώσουμε απλά ένα τάμπλετ. Θα πρέπει να αποκτούν την εμπειρία ούτω ώστε, ε, ώστε να μάθουν την αποτελεσματικότητα των ψηφιακών δεξιοτήτων διότι σε περίπτωση που δεν καταλαβαίνει μονάχα αν το καταλάβει αυτό θα μπορέσει να έχει κριτική σκέψη και να είναι δημιουργικό στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών και να μπορεί να ανταποκριθεί σε μια σύγχρονη τεχνολογία και τον ψηφιακό κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει συνεχώ να επικεντρώμαστε σε αυτό ούτω ώστε σταδιακά να μπορούν τα παιδιά να μαθαίνουν την ενασχόληση με την ψηφιακή τεχνολογία και ταυτόχρονα να έχουν την κριτική σκέψη τους ώστε να κάνουν ασφαλή περιήγηση στο ίντερνετ και να υπάρχουν ξεκάθαροι στόχοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να ε, παραδώσουμε ψηφιακές δεξιότητες και στους ηλικιωμένους ανθρώπους. Ε, η Ζαμπίνε το ανέφερε αυτό. Θα πρέπει να γίνει το μεγάλο άλμα ε, στο, όσον αφορά την πρόοδρο των μαθητευόμενων Γι' αυτό το λόγο λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στην ημεράσια διάταξη και θα πρέπει επιτέλους να ακολουθήσουν και πράξεις. Έχουμε πει αρκετά λόγια, όμως ε, περιμένω και από την Κομισιόν να υπάρχει ε, έργο το οποίο να υποστηρίζει, διότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για τα κράτη-μέλη και γι' αυτό το λόγο και τα ίδια τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνε τους και να δεσμευτούν ακόμα πιο πολύ πάνω σε αυτό το θέμα και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη ενασχόληση πάνω σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ε, ευχαριστώ πολύ η Γιάννα Τσικνάντσκα είναι εδώ. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Μια και εργάζομαι με άτομα που έχουν προβλήματα υγείας, δεν θέλω να ρωτήσω κατά πόσο λαμβάνονται αυτές οι ιδιαιτερότητες υπόψη και επίσης η αναγνώριση των δεξιοτήτων, γιατί στην Σλοβακία δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αναγνώριση των δεξιοτήτων μας σε άλλα κράτη-μέλη ή αντίστροφα. Υπάρχει περίπτωση φοιτήτρια με διδακτορικό στην ψυχολογία σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο. της, ε, στη Σλοβακία όμως δεν έγινε δεκτή διότι δεν είχε πάρει το πτυχίο Masters. Δεν είχε αναγνωριστεί καλύτερα το πτυχίο αυτό και γι' αυτό θα ήθελα να μάθω τι είδους μέτρα μπορούμε να εξασφαλίσουμε για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Και τρίτον, θα ήθελα πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τις ε, ψηφιακές δεξιότητες στον ιδιωτικό τομέα. Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα αυτό. Καλώς. Ευχαριστώ κυρία Μακλάρκιν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ τους δύο επιτρόπους που ήρθαν να μας μιλήσουν στις ε, Επιτροπές Απασχόλησης και Εκπαίδευσης. Έχω εργαστεί πάνω σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και στα θέματα της αμοιβαίας ανταγνώρισης. Περιμένω λοιπόν να ακούσω τις δικές σας νέες ιδέες και ιδιαίτερα τα θέματα σχετικά με την αναθεώρηση του ε, πλαισίου του 2008 για την αμοιβαία αναγνώριση. Πώς μπορεί αυτό λοιπόν να βοηθήσει τους νέους στην Ευρώπη. Και ίσως μπορείτε να μας δώσετε κάποιες, κάποια παραδείγματα ε, των πορισμάτων της δημόσιας διαβούλευσης στην οποία έχετε προβεί. Γιατί θα θέλαμε να συμπεριληφθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς σε αυτό το δημόσιο διάλογο και οι επιχειρήσεις, οι εργοδότες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τα ίδια. Επίσης γνωρίζω ότι η εκπαίδευση είναι αρμοδιότητα αποκλειστική των κρατών μελών. Όταν μιλούμε λοιπόν για εκπαίδευση, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνεται ε, αυτόνομα και χωριστά η δουλειά από το κάθε κράτος μέρος, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε στο πρώιμο δυνατόν, κατά το δυνατόν στάδιο συνεργασία, χωρίς να ζητούμε βέβαια πλήρη εναρμόνιση. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μας πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο προς την αναθεώρηση των οδηγιών και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, πώς σχεδιάζεται να επηρεάσετε σε αυτό το πιο πρώιμο στάδιο την διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Κύριε Αντλαμπάιωβα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους δύο επιτρόπους οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ικανότητες είναι κάτι το απαραίτητο και εγώ και άλλοι συνάδελφοι έχουμε δώσει αγώνα για αυτές πολλούς μήνες. Χρειάζεται να διευκρινιστούν θέματα στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης όπως επίσης και της πολλαπλότητας των ικανοτήτων σε πάρα πολλούς τομείς. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε ιδιαίτερα σε ορισμένα κρατημέλη, οι ανάγκες είναι υψηλότατες. Δεν χρειάζεται να καταστήσουμε κάθε Ευρωπαίο επιχειρηματία, αλλά είναι σαφές ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ε, ε, στοιχεία επιχειρηματικότητας. Χρειάζεται λοιπόν εδώ να ανταλλάξουμε γνώσεις και προτάσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν μιλάμε για ικανότητες, δεν θα πρέπει να τις βλέπουμε απομονωμένα, αλλά θα πρέπει να τις βλέπουμε πάντα συνδεδεμένες με την αγορά εργασίας. Θα πρέπει εδώ να, συν, ενισχύσουμε τον σύνδεσμο ανάμεσα στην απόκτηση των ικανοτήτων και στις ανάγκες της μελλοντικές της αγοράς εργασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή λοιπόν θα πρέπει να βοηθήσουμε στον καλύτερο συντονισμό των εκπαιδευτικών κέντρων, των σχολείων, των σχολών κτλ και έχουν οι μονάδες αυτές μάθηση, συζητήσει έτσι ώστε να μαζί με τα κράτη-μέλη και τις υπόλοιπες υπηρεσίες για να γνωρίζουν ποιες είναι οι μελλοντικές τους ανάγκες. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό και ακριβώς στα πλαίσια ιδιαίτερα της επαγγελματικής κατάρτισης οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές. Θα πρέπει επίσης ε, το θέμα της ε, διδασκαλίας των ικανοτήτων να καλύψει και τις ανάγκες των διδασκόντων. Ποιοι είναι αυτοί που θα διδάξουν τις ικανότητες ε, στους υπόλοιπους πολίτες. Αυτό είναι ένα ειδικότερο θέμα που θέλει απάντηση. Ευχαριστώ. Η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή είναι σημαντική και θέλω να ευχαριστήσω τους δύο επιτρόπους. Η συνάδελφος Μαρτίνα έκανε μια ξεκάθαρη δήλωση με την οποία συμφωνώ. Δυστυχώς ε, υπάρχει ένα θέμα το οποίο μέχρι τώρα δεν έχουμε εξετάσει. Το θέμα των ε, ε, του πλαισίου των ικανοτήτων του κοινοτικού είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο, αλλά δεν είναι όμως επαρκές. Έχουμε επίσης προβλήματα όταν ένας πολίτης πηγαίνει σε μία άλλη χώρα να αντιμετωπίζει τα θέματα της αγοράς εργασίας ακόμα πιο περίπλοκα λόγω της έλλειψης πολλές φορές επαρκών γλωσσικών γνώσεων σε χώρες όπως η Εσθονία, Λετωνία κτλ. υπάρχουν συγκεκριμένες γλωσσικές απαιτήσει και γλωσσικές ρυθμίσεις οι οποίες είναι ιδιαίτερως δεσμευτικές και πιεστικές. Θα πρέπει λοιπόν να μην απαιτούνται περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορέσει κανείς να λειτουργήσει σωστά επαγγελματικά. Γιατί αλλιώς αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν μια υπερβολή και καταχρηστική ρύθμιση στην ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων. Δυστυχώς οι ρυθμίσεις αυτές ε, που ισχύουν στα διάφορα κράτη-μέλη δεν σέβονται πάντα και δεν είναι πάντα συμβατές με την αρχή της αναλογικότητας. Οι δυνατότητες αμφισβήτησής τους υπάρχουν σήμερα μόνο σε δικαστικό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να δούμε ακριβώς τι γίνεται σε σχέση με την αγνώριση των ικανοτήτων και την αναγνώριση των γλωσσικών ικανοτήτων. Ε. Σας ευχαριστώ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πλέον η δυνατότητα για τους δύο επιτρόπους με πάρα πολύ σύντομο τρόπο να δώσουν ερωτήσεις, να απαντήσει συγγνώμη, σε όλες τις ερωτήσεις που προηγήθηκαν. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει έτσι κι αλλιώς για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Η κυρία Τάισεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε για τις πρώτες ερωτήσεις για την επιχειρηματικότητα τι μπορούμε να κάνουμε εμείς να διευκολύνουμε και να δώσουμε κίνητρα για την επιχειρηματικότητα. Η διερμηνία θα έλεγα του Κοινοβουλίου είναι άψογη και γι' αυτό παρασύρομαι και ομιλώ την Αγγλική. Τώρα θα αναγκαστώ να ομιλήσω όμως την Ολλανδική για να απαντήσω πληρέστερα. Σχετικά λοιπόν με τις ε, επιχειρηματικές γνώσεις και το πνεύμα της επιχειρηματικότητας, αυτό είναι πράγματι κάτι που πρέπει να ενισχύσουμε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το δούμε το θέμα σφαιρικά, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εργαστούμε σε όλα τα μέτωπα ταυτόχρονα. Θα πρέπει όλοι να έχουν τις αρμοδιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για να φέρουν εις πέρα στην δουλειά τους. Όταν μιλάμε για επιχειρηματικό πνεύμα, μιλάμε για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τα startups τα λεγόμενα οι πρωτοβουλίες υπάρχουν. Θέλουμε αυτό το πνεύμα της καινοτομίας να το μεταφέρουμε και να το εμφυσίσουμε σε όλους τους νέους. Δεν είναι εύκολο. Απαιτείται από όλους δημιουργικότητα, πρωτοβουλία και γνώση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Είναι δύσκολα θέματα. Θα πρέπει όλοι να κατανοήσουν ότι από τη μια μέρα στην άλλη δεν γεννιούνται νέοι επιχειρηματίες. Τώρα, άλλο θέμα, όταν μιλάμε για αυτούς που είναι άνω των 50 ετών, τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτον, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις ικανότητές τους έτσι ώστε να καταστούν απασχολήσιμοι. Την προηγούμενη εβδομάδα ήδη επισκεφθήκαμε την υπηρεσία για την ασφάλεια και την υγεία στους τόπους εργασίας. Ένα θέμα με το οποίο ασχολείται είναι ακριβώς η υγεία των εργαζομένων, ιδιαίτερα για τους προχωρημένης ηλικίας εργαζομένους, οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να ζήσουν εν πλήρη υγεία και μετά τη συνταξιοδότησή τους. Το θέμα της υγείας λοιπόν των εργαζομένων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παρακολουθήσουμε από πάρα πολύ κοντά, ιδιαίτερα για τους εργαζομένους άνω των 50 ετών γνωρίζουμε ότι οι πολίτες που, έχουν, άνω που είναι άνω των 50 ετών αντιμετωπίζουν δυσκολίες για να μπουν στην αγορά εργασίας και γι' αυτό δεν θα πρέπει να βγαίνουν από την αγορά εργασίας. Κάποιος ο οποίος έχει την εμπειρία των 50 ετών είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να προσφέρει πολλά στην επιχείρηση. Τώρα, για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, πώς περνά κανείς από το σχολείο στην δουλειά. Αυτό είναι δύσκολο σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ε, μία από τις καλύτερες μεθόδους για να διευκολυνθεί αυτό το πέρασμα ε, είναι η λεγόμενη διοική εκμάθηση, δηλαδή να προσπαθεί κανείς να σπουδάζει εν περιπτώσει, στα κέντρα εκπαίδευσης, αλλά να προσπαθεί να λαμβάνει στοιχεία εκπαιδευτικά και στους τόπους εργασίας. Αυτό θα τον διευκολύνει στο να κατανοήσει τις ανάγκες στον τομέα της εργασίας. Πολλοί από εσάς αναφερθήκατε στις ανάγκες των διδασκόντων που διδάσκουν αυτές τις ικανότητες. Ε, και αυτό είναι δύσκολο θέμα. Θα πρέπει να υπάρχει μια επαφή των εργαζομένων αυτών με την πραγματική οικονομία, με την πραγματική ζωή, με τις οικονομικές δραστηριότητες, τις βιομηχανίες κτλ. για να ξέρουν τι ε, απαιτείται από τους μαθητές τους. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει τεθεί νομίζω σε μένα είναι το πώς θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες ε, στον τομέα ιδιαίτερα της πρόσβασης σε προγράμματα κατάρτισης. Ήδη από το μήνα Μάρτιο ξεκινήσαμε μια μεγάλη συζήτηση σε αυτό το οποίο ονομάζουμε Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Μία από τις τρεις κατευθυντήριες γραμμές του συγκεκριμένου αυτού πυλώνα είναι ακριβώς ε, η ισότητα ευκαιριών. Στο εσωτερικό επίσης του πυλώνα υπάρχει φυσικά και η διάσταση η σχετική με τις ε, ε, ικανότητες. Το να έχει κανείς συγκεκριμένες ικανότητες είναι βασικός παράγων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Δεν είναι ο μοναδικός αλλά ο βασικός. Οι γυναίκες έχουν επίσης και το θέμα του φύλου το οποίο μπορεί μερικές φορές να δημιουργήσει προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν την διάσταση του φύλου να αντιλαμβάνουμε υπόψη σε όλους τους τομείς. Για τις ψηφιακές γνώσεις, επίσης ε, ε, σημαντικό πράγμα, θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε όλα τα συστήματα κατάρτισης. Στις σημερινές θέσεις απασχόλησης και πόσο μάλλον τις αυριανές, το 80% των εργαζομένων θα πρέπει με τον ένα τρόπο ή τον άλλο να χρησιμοποιούν ψηφιακού τύπου γνώσεις. Ακόμα και όταν εργάζεται κάποιος σαν ξυλουργός σε μια οικοδομή πρέπει να είναι ικανός στο να χειρίζεται ένα υπολογιστή για τεχνικούς λόγους. Θα πρέπει λοιπόν οι μελλοντικοί εργαζόμενοι να μπορέσουν να αποκτούν θεμέλια ε, στον τομέα της ε, χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε συντονιστικά εμείς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι πράγματι μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αντιμάχεται την αρχή της επικουρικότητας. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι τα τρία θεσμικά όργανα δεν έχουν διακανονιστικές και εναρμονιστικές δυνατότητες και αρμοδιότητες. Αυτό μπορούν να το κάνουν τα κράτη-μέλη. Ε, τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα εδώ, σεβόμεθα την αρχή της επικουρικότητας. Οι τοπικές, περιφερειακές, εθνικές αρχές είναι οι κατεξοχήν υπεύθυνε για τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Μπορούμε όμως να συνδράμουμε ε, τις χώρες να βελτιώσουν τα προγράμματα αυτά, να ανταλλάξουν πρακτικές, να λειτουργήσουμε συντονιστικά με λίγα λόγια και έτσι μπορούμε να ενισχύσουμε τις διαδικασίες αυτές μέσω ακριβώς των προτάσεων. Ανταλλαγή των χρηστών πρακτικών λοιπόν και εδώ μπορεί να βοηθήσει και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και με τις συστάσεις σαν χώρα νομίζω ότι μπορούμε να επιμείνουμε εκεί όπου υπάρχουν ανάγκες για την πρόσκληση ικανοτήτων που θα καταστήσουν την επαγγελματική ιδιαίτερα κατάρτιση πιο σημαντικό ρόλο. Ήδη έχουμε δώσει τέτοιου είδους συστάσεις σε 15 χώρες μέλη. Οι κοινωνική εταίροι επίσης θα πρέπει να έχουν λόγο Νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτό το πακέτο των ικανοτήτων. Μπορούμε επίσης να στηρίξουμε οικονομικά κάποια προγράμματα τέτοια, να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν στους στόχους αυτούς τους οποίους θεωρούμε χρήσιμους για να δώσουμε ένα μέλλον στους νέους και δυνατότητες εργασίας, να καταστήσουμε τους νέους Απασχολήσιμος. Η λέξη δεν είναι ωραία, αλλά παρόλα αυτά είναι σημαντική λέξη. Ε, στο παρελθόν τέτοιες λέξεις τις θεωρούσαμε αδόκιμες, ε, τώρα όμως τις χρησιμοποιούμε συνεχώς. Πρέπει να καταστήσουμε τους νέους όχι μόνο ικανούς να βρουν μια θέση εργασίας, αλλά να παραμείνουν στην αγορά εργασίας και να μην αναγκαστούν να αποκολληθούν από αυτή και να μπουν στο περιθώριο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχω άλλες ερωτήσεις. Α, για τους εργοδότες. Φυσικά και οι εργοδότες πρέπει να συμμετέχουν. Η εργοδοσία έχει συγκεκριμένες ευθύνες και θα πρέπει να είναι σε επαφή και με τον κλάδο της κατάρκησης εκπαίδευσης. Αυτά τα αποφασίζουν πώς θα γίνουν τα κράτη-μέλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εμείς φέρνουμε σε επαφή τους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή τους εργαζομένους, τα συνδικάτα, τους εργοδότε και να διευκρινίζουν εκεί τις αρμοδιότητες του καθενός. Έτσι, <clears throat> οι κοινωνικοί εταίροι <clears throat> θα αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες. Έχουμε άλλωστε υπογράψει συμβάσεις με ε, οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Εργοδοσίας για την λεγόμενη Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Κατάρτιση η ευρωπαϊκή εργοδοσία έχει αναλάβει την υποχρέωση να δημιουργήσει θέσεις υψηλής ποιότητας. Το να μιλάμε για διοικής μορφής κατάρτιση, δηλαδή και στο σχολείο και στην δουλειά. Αυτό θεωρητικά ακούγεται σωστά, αλλά θα πρέπει όμως η δουλειά στην οποία θα καταλήγει η θέση απασχόλησης να είναι αξιοπρεπής και χρήσιμη. Πρέπει λοιπόν στα πλαίσια αυτής τη συμμαχίας για την κατάρτιση και την απασχόληση ε, όπως είπα κάναμε μια σύμβαση με, το, με την οργάνωση της Ευρωπαϊκής Εργοδοσίας και επίσης το ίδιο έγινε και στα πλαίσια της πρωτοβουλίας για τους νέους. Τώρα για τις γλωσσικές απαιτήσει. Είναι σημαντικό αυτό που είπατε. Φυσικά οι νέοι πρέπει να ομιλούν ξένες γλώσσες για να συμμετέχουν στην ε, δουλειά, ε, στην, στο χώρο δουλειά, στη χώρα που μένουν κτλ αλλά από την άλλη για λόγους προστατευτισμού δεν θα πρέπει να επιβάλλονται απίστευτα υψηλού επίπεδου γλωσσικά κριτήρια. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ που ε, περιοριστήκατε στο χρόνο που σας αναλογεί και η συνεισφορά σας ήταν πάρα πολύ καλή και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Επιτρόμο του Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα είμαι πιο σύντομος, το ελπίζω τουλάχιστον, διότι η Επίτρομος Τάισεν ε, έδωσε πάρα πολύ καλές απαντήσεις με τις οποίες συμφωνώ, οπότε για μένα έμεινε το εύκολο κομμάτι. Αρχικά, οι δεξιότητες, η απασχολησιμότητα δεν είναι μονάχα οικονομική ηθικοί όροι και κατηγορίες, είναι και κοινωνικοί όροι και κατηγορίες, διότι υπάρχουν ξεκάθαρες αποδείξεις ε, για τον συσχετισμό μεταξύ των κοινωνικών οικονοτήτων και υποβάθρου αλλά και την αποσχολησιμότητα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όταν μιλάμε για παράδειγμα για την επιχειρηματικότητα το ζήτημα δεν αφορά μονάχα το να διδάξουμε πώς ε, διευθύνεις μια εταιρεία, πώς ε, έχεις οικονομικές γνώσεις κτλ. Για μένα η επιχειρηματικότητα αφορά το να είσαι αυτόνομος, ανεξάρτητος πολίτης, πώς μπορείς να παίρνεις αποφάσεις σχετικές ε, για την ε, κοινωνία, για τις ε, καριέρες και το πώς να δημιουργήσεις μια αρμονία μεταξύ του συμφερόντος του μεμονωμένου ατόμου και της κοινωνίας. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι όταν μιλούμε για την επιχειρηματικότητα και την εκπαίδευση, Πρόκειται για μια οριζόντια δεξιότητα και το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να διδάσκει τις βασικές ικανότητες επιχειρηματικότητας, το να σκέφτεσαι υπεύθυνα, πώς να συνεργάζεσαι με μια κοινωνία, πώς να επιτύχει συμφωνία, πώς να εναρμονίσεις ε, διαφορετικές ε, προτάσεις. Ε, θα θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη στο να δημιουργήσουν τα στοιχεία ε, της επιχειρηματικότητας και να τα ενσωματώσουν στα εκπαιδευτικά συστήματα. Θα πρέπει να τα βοηθήσουμε να διδάξουν στοιχεία τα οποία αφορούν την οικονομική, πολιτισμική πλευρά της επιχειρηματικότητας, ταυτόχρονα όμως να τους ε, δείξουμε πώς να καλέσουν ε, στα σχολεία ε, πρότυπα της κοινωνίας, επιχειρηματικά πρότυπα, ούτω ώστε να δώσουν κάποιες μαρτυρίες σχετικά με τη δουλειά που κάνουν και τις ικανότητες που έπρεπε να έχουν για να μπορέσουν να είναι επιτυχημένοι είναι ε, μια πολύπλευρη δουλειά αυτή ε, και γι' αυτό το λόγο θα θέλαμε να δώσουμε την απαραίτητη βοήθεια για την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων στο μέλλον. Τώρα όσον αφορά τις ψηφιακές ικανότητες, ναι, έχουμε σημαντικά δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι το 70% των ε, διδασκόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζουν τη σημασία των, των ψηφιακών δεξιοτήτων στη σύγχρονη ζωή. Ταυτόχρονα όμως σε, σε σχολεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις το 25% των μαθητών διδάσκονται από ε, δασκάλους που είναι αρκετά καλά καταρτισμένοι στη ψηφιακή τεχνολογία. Οπότε θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στην εκπαίδευση των δασκάλων. Θα πρέπει πρώτα να ε, βοηθήσουμε αυτούς για να μπορέσουν αυτοί στη συνέχεια να διδάσκουν τους μαθητές οι οποίοι πολλές φορές έχουν καλύτερες ψηφιακές ικανότητες από ότι οι ίδιοι οι δάσκαλοι μέσα στην τάξη. Πρέπει λοιπόν να τους δώσουμε περισσότερες δυνατότητες, τους δασκάλους εννοώ για να μπορέσουν να προφτάσουν ε, σε μερικές περιπτώσεις τους μαθητές τους. Ένα από τα σημαντικά στοιχεία ε, του εκπαιδευτικού ε, μέρους του θεματολογίου είναι η εκπαίδευση των δασκάλων διότι θα πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε για να τοποκριθούν στις πιο σύγχρονες δεξιότητες. Τώρα όσον αφορά την επικουρικότητα Συμφωνώ με την Επίτροπο Τάισεν ότι μπορούμε να κάνουμε ε, πολλά και μπορούμε να δημιουργήσουμε μια διαφορά όσον αφορά την επιρροή στα κράτη-μέλη. Μέχρι στιγμής ε, θα δεν έχει επιτευχθεί μια απόλυτη συμφωνία, όμως ε, νομίζω ότι δεν πρόκειται να επιτευχθεί χωρίς ε, την υποστήριξη των κρατών μαλλών. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη συμφωνία, θα πρέπει να τα επηρεάσουμε και νομίζω ότι είναι σημαντικό ούτως ώστε να υπάρχει προωθηθεί καλύτερα το θεματολόγιο και από την άλλη ε, μπορούμε να οργανώσουμε ε, ανταλλαγή ιδεών, ε, workshop, καλύτερες πρακτικές ούτω ώστε να μπορέσουμε να επηρεάσουμε τα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, αυτή την περίοδο κάνω την αναφορά της πολιτικής Our Education και έχω ένα πολύ καλό feedback ε, από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πάνω σε αυτό το θέμα και οι ενδιαφερόμενοι ε, καθώς επίσης και η αγορά εργασίας έχουν στείλει αναφορές οι οποίες δείχνουν ότι θα πρέπει να, ε, βελτιώσουμε ε, τα επίπεδα απασχολησιμότητας, ε, θα πρέπει να φέρουμε την ακαδημαϊκή κοινότητα και την αγορά εργασίας ούτως ώστε να, να υπάρξει περισσότερη υποστήριξη όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση για τα πανεπιστήματα, για πανεπιστήμια για να μπορέσουν να προσαρμόσουν τα μαθήματά τους ούτω ώστε να γίνουν πιο πρακτικά ή τουλάχιστον να αναπτύξουν το πρακτικό κομμάτι πέραν του θεωρητικού. Έχουμε λοιπόν, θεωρώ, καλά αποτελέσματα σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα αναλάβει η πρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού, κυρία Κώστα. Ευχαριστώ. Και τώρα θα ακούσουμε άλλους συναδέλφους για το δεύτερο γύρο. Υπενθυμίζω ότι πρέπει οι ερωτήσεις σας να περιορίζονται στο 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα για τους βουλευτές και το πολύ σύνολο για τους δύο επιτρόπους στα 10 λεπτά οι απαντήσεις. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, έτσι ώστε να επιτρέψουμε μετά να δεξαχθεί και τρίτος γύρος ρωταπαντήσεων. Η κυρία Κούνεβα, παρακαλώ, από την ΚΟΕ. Απασχόληση. Έχετε το λόγο. Όσο και αν βελτιωθούν οι δεξιότητε, δεν αρκούν για να μειωθεί η ανεργία. Το γνωρίζουν πολύ καλά 25 εκατομμύρια άνεργοι. Οι έρευνε δείχνουν στην Ευρώπη ότι 6 άνεργοι αντιστοιχούν σε μια θέση εργασία. Ενώ το 2011 σε Ισπανία και Ελλάδα μια θέση αντιστοιχή και σε 20 ανέργους. Εάν επιμένουμε ότι θα λύσουμε το θέμα της ανεργίας δίνοντας προτεραιότητα στις δεξιότητες των ανέργων, είναι σαν να πιστεύουμε ότι για την ανεργία φταίνει οι άνεργοι. Χρειάζονται περισσότερες θέσει εργασία. Και αυτό δεν βλέπουμε πώς θα γίνει όταν δεν είναι στι προτεραιότητε τη Επιτροπή η δημιουργία θέσεων εργασία ω στο προσχέδιο των πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που δόθηκε προ διαβούλευση από την Επίτροπη Τίσεν η Κομισιόν πιστεύει ότι η βελτίωση της αντίστοιχη των δεξιοτήτων με την αγορά εργασία θα βελτιώσει, όπω λέει την αποσχολησιμότητα και θα πιάσουμε το στόχο ώστε το 2020 το 75% του εργάσιμου πληθυσμού θα έχει εργασία. Μα σε πολλές χώρες έχουμε πολύ καταρτισμένους άνεργους με αποτέλεσμα εκατοντάδε χιλιάδες να μεταναστεύουν στη Γερμανία και αλλού. Ποιο άνεργο το ΟΜΑ όταν έξω από την πόρτα περιμένουν χιλιάδες άνεργοι να ζητήσει από τον εργοδότη χρόνο κατάρτισης και βελτίωση των δεξιοτήτων. Η ερώτηση, τι τα κάνουν οι αυτό οι ενώσει των εργοδοτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χοντής παρακαλώ από την Επιτροπή Πολιτισμού Κουβά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των δύο επιτρόπων και αρκετές από τις απαντήσεις που έδωσαν μέχρι τα τώρα. Θέλω να πω ότι ποιος αντιλέγει ότι χρειάζεται καλλιέργεια των δεξιοτήτων, επικαιροποίηση των ικανοτήτων. Όμως πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν είναι και ικανή συνθήκη για να αντιμετωπίσει ή να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πρώτη ερώτηση λοιπόν έχει το χαρακτήρα ποιο πρόβλημα έχει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε μέσω της αναγκαίας αυτής της διαδικασίας. Είναι το πρόβλημα της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας που όπως λένε τα κείμενα δεν έχουμε και έχει έλλειψη εργατικών χεριών. Είναι το πρόβλημα της ανεργίας που είναι οξύτατο, έχουν αναφερθεί τα στοιχεία της ανεργίας ιδιαίτερα των νέων, ιδιαίτερα στην πατρίδα μου την Ελλάδα είναι ένα γενικότερο δικαίωμα, σωστά χαρακτηρίστηκε δημοκρατικό δικαίωμα που πρέπει να παρέχει εκπαίδευση ανεξάρτητα από κοινωνικέ αντιθέσει. Ποιο πρόβλημα θα λύσουμε. Πάντω όχι τη ανεργία. Δεύτερο, ε, λέτε και έχω παρακολουθήσει και την ε, προτεραιότητα τη Επιτροπή και το προηγούμενο χρόνο από άλλε θέσει. Είναι προτεραιότητα τη επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Αν πάλι αναποθέτουμε τα ζητήματα αυτά και βάζουμε όλο και πιο πολύ τι απαιτήσει τη αγορά στην εκπαίδευση, δεν θα το λύσουμε. Και το τελευταίο ερώτημα που συμπυκνώνει τι αντιφάσει το έθιξε και η συναδέλφισσα. Γιατί έχουμε διαρροή εγκεφάλων από τι χώρε του Νότου, πώ το αξιολογείτε, πού οφείλεται, πώ θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, ποιον ωφελεί ή πρέπει να υπάρχει για να λυθούν άλλα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, please. I invite to respect the... Ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να σας περιορίζω το χρόνο, αλλιώς δεν θα έχουμε αρκετό χρόνο όλοι οι συνάδελφοι. Λάμπερτς, παρακαλώ, η κυρία Λάμπερτς από τους Πράσινους, Επιτροπή Απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι περιμένουμε, νομίζω, το θεματολόγιο για τις νέες δεξιότητες. Συζητήσαμε σήμερα κάποιες βασικές Δεξιότητε απαραίτητες, βεβαίως ε, να μπορεί κανείς να γράφει, να διαβάζει, να κάνει βασικούς υπολογισμούς, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και το πλαίσιο με στο οποίο εργάζεται ο καθής και γι' αυτό θα περάσω στην έκθεση απασχόληση των πρασίνων. Την πράσινη έκθεση απασχόληση, συγγνώμη, που εγκρίθηκε το προηγούμενο Ιούλιο. Σε έναν βαθμό αναφερόταν και στο πώς μπορεί να μπει κανείς στην αγορά εργασίας, θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, αηφορία του περιβάλλοντος, την αποτελεσματική χρήση των πόρων, την χρήση των πόρων κατά τρόπο ορθολογικό. Αυτό ως γενικές δεξιότητες. Τι έχετε να πείτε, γι' αυτό δεν είπατε κουβέντα μέχρι τώρα. Και επίσης, οι βασικές δεξιότητες που μπορούν να αναπροσαρμόζονται όπως βέβαια η τεχνολογία, όπως ε, μηχανολογικές ή μαθηματικού τύπου δεξιότητες, έχουν ε, σαν χαρακτηριστικό ένα μεγάλο χάσμα στις γενναίες. Αυτό πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Είναι πολλές οι επιτροπές του Κοινοβουλίου που έχουν ένσκυψει το θέμα αυτό και δεν βλέπουμε λύση ακόμα. Επίσης, σε σχέση με τους εμπλεκόμενους φορείς που έθιξε και η κυρία Μακλάρκιν, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές τι ρόλο θα διαδραματίσουν γιατί θεωρείται ότι και αυτές μπορούν να έχουν ένα σημαντικό, ε, μια σημαντική και δυναμική συμβολή στο θεματολόγιο για τις Ευχαριστώ. Jill Πράσινη, Επιτροπή Πολιτισμού. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ την Ουαλία του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχουμε μια πολύ καλή εμπειρία από πρόγραμμα δεξιοτήτων που χρηματοδότησε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το οποίο ε, ωφέλησε ιδιαίτερα τους εργοδότες. Τους βοήθησε να στοχεύσουν πολύ πιο αποτελεσματικά την, ε, ε, τους σπόρους για την κατάρτιση και να εντοπίσουν τις ανάγκες σε κατάρτιση και σε μαθητεία βεβαίως πέραν του περιεχομένου, σε νέους ανθρώπους προς τους θέσεις εργασίας. Από τη μελέτη αυτή προκύπτει ξεκάθαρα ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις ο μικρής κλίμακας εργοδότης δηλαδή ήταν και πιο αποτελεσματικός στην αξιοποίηση του προγράμματος αλλά και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ε, χάρη ιδιαίτερα στην μαθητεία. Ερωτώ λοιπόν εάν αυτό μπορεί να είναι ένας ιδιαίτερο παράγον περισσότερο παρά στόχο ε, στο θεματολόγιο της δεξιότητας. Πρέπει να κοιτάξουμε το ρόλο των μικρών και πολύ μικρών μερικές φορές εργοδοτών και επίση τα όσα είπε η Jean Lambert, η συνάδελφο εδώ. Οι δημόσιε αρχέ, τοπικέ και περιφερειακέ ιδιαίτερα, ε, τι ρόλο μπορούν να διδραματίσουν, γιατί αυτές αποτελέσουν και τους κινητήριους μοχλούς, στη τελευταία ανάλυση. Ευχαριστώ. Λάουρα Τζέα, απασχόληση, ομάδα EFTD. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους επιτρόπους ε, οι οποίοι μας έδωσαν τελικά ένα πανόραμα ίσως όχι πολύ συγκεκριμένο της κατάστασης. Εγώ ξεκινώ από μια προϋπόθεση η οποία δεν είναι αμφισβητήσιμη. Στην ηλική φτώχεια ανταποκρίνεται και η πνευματική, πολιτιστική καλύτερα, συγγνώμη, φτώχεια. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό των γνώσεων, θα πρέπει να εξηγιάνουμε καταρχάς και να αντιμετωπίσουμε το, το πρόβλημα της φτώχειας είναι κάτι το οποίο δυστυχώς μαστίζει πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Θα συμφωνήσω και με τον συνάδελφο Κάζα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα τρομερό πρόβλημα, το πρόβλημα της ανεργίας μακράς διάρκειας και αυτό δημιουργεί προβλήματα και στον τομέα του αλφαβητισμού και πέραν αυτό. Ε, απαιτείται λοιπόν ότι πρέπει να βοηθήσουμε την ανάκτηση ικανοτήτων και να θέσω και μία ερώτηση. Αναφερθήκατε στην απασχολησιμότητα και την απασχόληση. Είναι δύο πράγματα, είναι ένα πράγμα. Εγώ έχω την αίσθηση ότι έχουμε να κάνουμε με δύο αντιλήψεις, οι οποίες μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά έχουν και τρομερές διαφορές μεταξύ τους. Ε, να χρησιμοποιεί ο καθένας τις αρμοδιότητες του ή μήπως να δουλεύει έτσι κι αλλιώς ανεξαρτήτως του τι δουλειά κάνει. Εγώ τα 15 χρόνια που έχω δουλέψει μέχρι τώρα ε, είχα την δυνατότητα να χρησιμοποιήσω γνώσεις υψηλού επίπεδου, αλλά μήπως θα έπρεπε να προσπαθήσω να μάθω και άλλα πράγματα. Ένα άλλο πράγμα είναι οι νεοφυείς επιχειρήσεις, τα start-ups ε, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να πουλήσουμε σαν μαγική λύση. Του, ε, Ευχαριστώ, Ντομινίκ Μαρτά. Ευρω... Ε, ΕΝΦ και απασχόληση. Ευχαριστώ. Ωραία πράγματα άκουσα. Πολύ ωραία πράγματα κοινή λογική. Να μάθει κανεί να γράφει, να διαβάζει, να μετράει, ψηφιακέ δεξιότητες για τους νέους μας, επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση, διαβίου μάθηση με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, αξιοποίηση των εμπειριών ε, της επιχειρηματικότητας, παρακολούθηση την εξέλιξη των, δεξι, των δεξιοτήτων ε, και βέβαια δεν αναφέρθηκε αλλά πιστοποίηση της κτήση. Ε, των εμπειριών και δεξιδιτών. Πολύ ωραία όλα αυτά για να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα, όπως υπόθηκε πρώτον. Δεύτερον, για να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αισθάνομαι ε, σε πολύ δύσκολη θέση, αισθάνομαι τρόμο και ως και φόβο, γιατί έχω την εντύπωση ότι συμμετέχω σε ένα συνέδριο αναπτυσσομένων κρατών στη δεκαετία του 70 σαν να έχουμε κάνει ένα άλμα προς τα πίσω, ένα τεράστιο άλμα προς τα πίσω. Αυτά τα προβλήματα είχαν αυτοί οι λαοί ε, στη δεκαετία του 70. Ή αλλιώς με στην Επιτροπή Απασχόλησης Πολιτισμού Παιδείας στις 18 Απριλίου του 2016 με νούμερα απίστευτα. 20% 1 πέμπτο των ε, νηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναλφάβητη και αντίστοιχα 9 εκατομμύρια φτωχοί. Είμαστε η έκτη δύναμη στον κόσμο. Ε, και είμαστε έκτη σε σειρά επίση σε αναλφαβητισμό. Δηλαδή, όσο περισσότερη Ευρώπη υπάρχει, τόσο χειρότερα πάντα πράγματα. Και κυρία Τάισεν, για να τελειώνω, ε, θέλουμε απασχολήσιμου πολίτε να φτιάξουμε πολύ ωραία και μπράβο μα, αλλά κυρία Τάισεν, αυτό μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν υπάρχουν και οι επιχειρήσει για να απασχολούν του απασχολήσιμου εργαζομένου και η Ευρώπη δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να τι καταστρέφει τι επιχειρήσει. Ευχαριστώ. Dominic Enf, πολιτισμός. Κυρία και κύριε Επίτροπε, αντιλήφθη πολύ καλά ότι η προσεχή δραστηριότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, απασχόληση θα βελτιώσει την απασχολησιμότητα των νέων, ζωτική ε, προτεραιότητα με δεδομένη την ενεργία έω και 50% στην Ελλάδα, παραδείγματι των νέων, και σε άλλε χώρε αύξηση ενεργείας από την εκείνη τη λειτουργία τη πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, όπω συνέβη στη Γαλλία. Οι εκπαιδευτικοί έχουν κρούν στον κόδωνα του κινδύνου για τους κινδύνου της πρωτοβουλία, σας σε σχέση με την, με την εκπαίδευση και κυρίως τη χρηματοδότηση που θα στηρίζεται στις επιδόσεις των δημοσίων σχολών, ΕΦΠ όπως ονομάζονται, και μπορεί να είναι βεβαίω απαραίτητο να αναπτυχθεί ο σύνδεσμος με την επιχειρηματική δραστηριότητα και κυρίως τη μικρομεσαία επιχείρηση. Ωστόσο, η σχολική πορεία, η εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει και σε ανατροπή της ισότητα των ευκαιριών όπως επισημαίνει το UCU, ε, το Βρετανικό Σωματείο Διδασκόντων, υπάρχει κίνδυνος εάν, άνθρω... εάν φοιτητέ, μαθητέ οι οποίοι έχουν πνευματικές δυσκολίες εγγράφονται σε σχολές μπορεί να μην γίνονται δεκτοί, γιατί θα θεωρηθεί από τη σχολή ότι μπορεί αυτό να αυξήσει το κόστος. Τη λειτουργία τη σχολή. Πώ λοιπόν κύριε Ρεναβασίτης σκοπεύετε να κάνετε την ποιοτική και όχι μόνο την ποσοτική αξιολόγηση τη λειτουργία των σχολών. Υπάρχει δυνατότητα με την εκπαίδευση και τα νέα μέτρα όπω το ευρωπαϊκό πλαίσιο επιστοποίηση, να ε, υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη. Και τρίτη ερώτηση αντίστοιχη με αυτή του συναδέλφου, δηλαδή στο θεματολόγιο αυτό η απόκτηση των θεμελιωδών δεξιοτήτων. Παρακαλώ να ολοκληρώνετε λέει η κυρία Κώστα. Καλώ ευχαριστώ and 50, sorry. Now, now Πέντε λεπτά τώρα. Έκαστος Επίτροπος, παρακαλώ. Και μετά θα έχουμε έναν τρίτο γύρο. Ενημερώνω τους συναδέλφους. Μετά τις δύο αυτές λεπτές παρεμβάσεις θα γίνει ένας τρίτος γύρος για τους συναδέλφους, όποιος ενδιαφέρεται για ένα λεπτό μόνο. Ποιο θέλει να ξεκινήσει. Θέλετε εσείς κύριε Ναυρατσίτς. Καλώς. Μια-δυο προτάσεις μόνο. Απασχολησιμότητα και απασχόληση. Φυσικά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η απασχολησιμότητα είναι μια ευκαιρία, ενώ η απασχόληση είναι ένα γεγονός. Η εκπαίδευση συνεισφέρει στην απασχολησιμότητα αλλά είναι πολύ δύσκολο να συνεισφέρει στην απασχόληση. Τα σχολεία είναι βέβαια και εργοδότες, αλλά στόχος τους είναι να δώσουν γνώσεις στους πολίτες να έχουν δυνατότητες για την αγορά εργασίας. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε τη διάκριση, να ενισχύσουμε τα σχολεία έτσι ώστε οι διδάσκοντες να εμφυσίσουν στους νέους πολίτες τις ικανότητες που απαιτούνται για να δουλέψουν και θα συμφωνήσω εδώ με την κυρία Τάισεν. Νομίζω ότι και το δικό μου χαρτοφυλάκιο μπορεί να προσφέρει εδώ, αν και της κυρίας Τάισεν περισσότερα. Τώρα για τη χρηματοδότηση των νέων που αντιμετωπίζουν θέματα που μειονεκτούν και τα λοιπά έτσι ώστε να προετοιμαστούν για την αγορά εργασία. Κοιτάξτε, στο Erasmus Plus υπάρχουν μέτρα καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Πρέπει να καταστήσουμε τα προγράμματα Erasmus Plus πιο προσβάσιμα στις κατηγορίες νέων που έχουν περισσότερα θέματα. Σεβόμενοι πάντα την αρχή της επικουρικότητας βέβαια. Δεν υπάρχει δηλαδή άμεση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα εκπαιδευτικά συστήματα. Πρέπει όμως να βοηθήσουμε τους νέους που έχουν ε, κάποια μειονεκτήματα, που αντιμετωπίζουν μειονεκτήματα. Η κυρία Τάισεν, η Επίτροπος Τάισεν έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι ιδιαίτερα σύντομη. Είναι σαφές ότι με τις σωστές ικανότητες και με συμμετοχή ενεργή και δραστήρια δεν γεννάει κανείς θέσεις απασχόλησης απαιτείται ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, απαιτείται μια καλύτερη μακροοικονομική πολιτική. Και εδώ το στρατηγικό πρόγραμμα επενδύσεων του Πρόεδρου Γιούνκερ μπορεί να βοηθήσει. Έτσι θα προσελκύσουμε και ιδιώτες επενδυτές έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες στον τομέα της απασχόλησης. Απ' την άλλη όμως έχουμε ανάγκη από πολιτικές στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν μέρος στη συγκεκριμένη αγορά, βελτιώνοντας λοιπόν τις ικανότητές τους, τους καθιστούμε πιο αντίστοιχους με τις ανάγκες της αγοράς. Το πρόγραμμά μας στον τομέα αυτό των ε, ικανοτήτων και αρμοδιοτήτων έχει σαν στόχο φυσικά και την ανάπτυξη, δεν το κρύβουμε αυτό. Ξέρετε ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία έχει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα ακόμα και δημογραφικού τύπου. Πρέπει λοιπόν να καλύψουμε τις ανάγκες των πολιτών. Έχει σημασία λοιπόν να καλύψουμε τις ανάγκες των πολιτών. Ε, τώρα για την φυγή των εγκεφάλων. Ε, να εκπαιδεύουμε φυσικά ανθρώπους οι οποίοι θα φύγουν κάποια στιγμή. Αυτό είναι ένας κίνδυνος. Απ' την άλλη η κινητικότητα είναι μια ευκαιρία. Η κινητικότητα είναι κυκλική όταν κάποιο δεν βρίσκει να δουλέψει σε ένα μέρος, ναι μεν πηγαίνει κάπου αλλού για να αναζητήσει θέση απασχόλησης, αλλά μαθαίνει εκεί που πάει και πολλέ φορές επανέρχεται στη χώρα εκκίνηση. Τώρα για τις πράσινε θέσεις απασχόλησης. Είναι σαφές ότι εδώ η περιφερειακή διάσταση και η τοπική διάσταση θα παίξει σημαντικό ρόλο. Όταν βλέπουμε τις γνώσεις που απαιτούνται για τις πράσινες θέσεις εργασίας, μένει πολλά να γίνουν. Είναι σαφές προς την Ευρώπη υπάρχουν λίγοι οι οποίοι έχουν τέτοιου είδους ικανότητες και δεν υπάρχει σφαιρικός τρόπος αντιμετώπισης των θεμάτων αυτών. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες λοιπόν των διαφόρων κοινοτήτων. Η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου έμεσα και σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο. Τώρα για την καταπολέμηση της φτώχειας και το πόσο συνδέεται με το θέμα των αρμοδιοτήτων. Κοιτάξτε, η φτώχεια απομακρύνει και αποκλείει τους πολίτες. Φυσικά η καταπολέμηση της φτώχειας θα πρέπει να γίνει σε όλα τα επίπεδα και γι' αυτό ακριβώς στις συστάσεις αναχώρα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο απευθύναμε συστάσεις προς πολλά κράτη-μέλη έτσι ώστε η σε ορισμένες χώρες να βελτιωθούν τα συστήματα υποδοχής ακόμα και των μικρών παιδιών. Το σύστημα πρέπει να λειτουργεί καλά από μικρή ηλικία, από τα, τους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία. Και πάρα πολλοί πολίτες σε πολλές χώρες έχουν προβλήματα να συνδυάσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα με την οικογενειακή ζωή δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους όπως θέλουν γιατί δεν έχουν τις απαραίτητες δομές ε, τις οποίες να χρησιμοποιήσουν για να μπορέσουν να δουλέψουν ελεύθερα. Πρέπει λοιπόν να ισορροπήσουμε με καλύτερο τρόπο την επαγγελματική ζωή με την οικογενειακή ζωή. Είναι βασικό αυτό όχι μόνο για τις γυναίκες αλλά κυρίως για τις γυναίκες, ιδιαίτερα των χαμηλών οικονομικών ε, στρωμάτων. Ο συνδυασμός αυτών των δύο, αν θέλετε, διαστάσεων είναι ιδιαιτέρως ε, δύσκολος. Τώρα για την ε, ανεργία μακράς διάρκειας. Ε, ίσως ε, να μην ε, μας είπατε ότι δεν ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με αυτό, μα ίσα ίσα εμείς ζητάμε εδώ και πολύ καιρό από τα κράτη-μέλη να κάνουν διαφορετικές τροποποιήσεις στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε οι άνεργοι, αυτοί οι μακροπρόθεσμα, μακροχρόνια άνεργοι να έχουν επαφές με την αγορά εργασίας και έτσι μόνο θα έχουν δυνατότητες να βρούνε μια δουλειά που να ανταποκρίνεται στην δική τους κατάσταση και ανάγκη. Αυτή η αντιμετώπιση είναι λειτουργική θα έλεγα, όχι γιατί την προτείνουμε εμείς, αλλά γιατί βασίζεται στην ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στις χώρες. Ξέρουμε τι δουλεύει, ξέρουμε τι δεν δουλεύει και προσπαθούμε να βρούμε τις σωστές λύσεις. σας ζητώ συγγνώμη. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στα μέλη, όμως ε, μας έχει μείνει λιγότερος χρόνος ε, από ό,τι ε, είχαμε προβλέψει και αυτό το λόγο κάθε βουλευτής θα έχει ένα λεπτό και στη συνέχεια πέντε λεπτά για τους ε, επιτρόπου. Έχουμε στη λίστα μέχρι στιγμή 11 ευρωβουλευτέ και αυτό το λόγο θα σα να περιοριστείτε στο ένα λεπτό διότι αλλιώ δεν πρόκειται να προλάβουμε. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Ασαρτέ από το ΕΠΠ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τέσσερα σημεία στο οποίο θα θέλω να ακούσω απαντήσει από του επιτρόπου. Το πρώτο αφορά την απόκτηση του βασικού βάθρου. Ανάγνωση, γραφή και ε, βασικοί υπολογισμοί, πώς μπορούμε να προωθήσουμε τις κατευθύνσεις αυτές για τα κράτη-μέλη για να υπάρχουν αυτές οι βάσεις, τις οποίες δεν μπορούν να προοδεύσουν οι άνθρωποι. Δεύτερον, πώς θέλετε, πώς σκοπεύετε να εξασφαλίσετε τη σύγκληση της ε, εκπαίδευσης που είναι χρόνος μακρός, της απασχόλησης που είναι χρόνος ε, μέσο και της ψηφιακής κατάρτισης που είναι χρόνος βραχής. Και αυτοί οι τρεις χρόνοι πρέπει να συγκλίνουν. Και τρίτον, ε, επικοινωνία. Επικοινωνία μεταξύ, όπως είπατε, των εκπαιδευτών που πιστεύουν ότι προσφέρουν τις κατάλληλες δεξιότητες και των επιχειρηματιών που έχουν την ε, αντίστροφη στάση και θεωρούν ότι δεν προσφέρονται επαρκείς δεξιότητες. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό για την ε, παιδεία, το καταφέραμε, αλλά για τις λοιπές καταρτήσεις. Και επίσης τα βιογραφικά του μέλλοντος πώς μπορούν να προβάλλουν δεξιότητες αντί για πτυχία περισσότερο. Από θεματικά επαγγελματικά πτυχία πρέπει να περάσουν σε εγκάρσιες δεξιότητες. Ευχαριστώ. Μαρία Ρενά, S&D. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρώτη ερώτηση αφορά την εκπαίδευση. Έχουμε τις έρευνες της Πίζας που δείχνουν σήμερα πως ε, ε, στην Ευρώπη το πρόβλημα παρουσιάζεται όχι ως προς, τις, ε, ως προς την αριστεία, αλλά ως προς την ισότητα, ως προς την ισότιμη πρόσβαση σε αυτές από το σχολικό σύστημα. Αυτό δεν το θίξατε καθόλου, τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν, ως προς την ισότιμη πρόσβαση και την ισονομία. Ε, δεξιότητε δεύτερον. Πολύ σωστά λέει η κυρία Τισένα ότι πρέπει να επενδύσουμε στι δεξιότητε. Δυστυχώ όμω από εμπειρία βλέπουμε ότι μπορούμε να επενδύουμε πολλά σε τομεί υψηλή ε, ένταση εργατικού δυναμικού όπω τον κατασκευαστικό τομέα που όμω λόγω των κοινωνικών προβλημάτων και παρά τι δεξιότητε οι άνθρωποι αυτοί μένουν άνεργοι γιατί δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί έναντι εργαζομένων που κοστίζουν 30 και 40% ακόμη φθηνότερα, προερχόμενοι από ευρωπαϊκά πάντα κράτη. Ερωτώ λοιπόν τι θα κάνετε γι' αυτό. Και τρίτη ερώτηση, για την ε, λιτότητα. Υπάρχουν προγράμματα λιτότητας τα οποία δεν επιτρέπουν επενδύσεις σε προγράμματα γνώσης της, ε, της του θα Αν δεν αλλάξουμε αυτά τα προγράμματα λιτότητας θα δούμε ανθρώπους που και σήμερα και αύριο και σε 20 χρόνια δεν θα έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες. Ευχαριστώ Σαντέρ Ελκ, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, απασχόληση. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να αναφερθώ σε δύο ζητήματα. Πρώτον, την κινητικότητα, γιατί θεωρώ πως πρέπει να καταβληθούν πολύ σοβαρές προσπάθειες για να διευκολυνθεί η κινητικότητα και κυρίως των μαθητευομένων. Υφίσταται μια σειρά εργαλείων όπως το Εργασμούς Plus, αλλά πολλές είναι και οι δυσκολίες στην πρόσβαση για τους μαθητευομένους σε αυτά τα μέσα είτε γιατί είναι πολύ νέοι, γιατί υπάρχουν προβλήματα στέγης, μεταφορών ε, ή και καθεστώτος του μαθητευομένου και ρωτώ αν υπάρχουν κάποιες λύσεις ε, προς την κατεύθυνση αυτή. Δεύτερον, κινητικότητα των ε, στελεχών επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών των ίδιων. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα μέσα του έρασμους προς όφελος των επιχειρηματιών. Και τρίτον, δυσκολίες σε ορισμένες ε, παραμεθορίους, όπου σημειώνεται ανταγωνισμός στη διεκδίκηση των δεξιοτήτων. Κάποια κράτη προσφέρουν εκπαίδευση σε συγκεκριμένε δεξιότητε, όπω επί παραδείγματι στην ορολογοποιία, ε, και στη συνέχεια κάποια άλλα κράτη είναι αυτά που απορροφούν το καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. Ευχαριστώ. World Cult. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο γρήγορα ερωτήματα. Το πρώτο αφορά ε, την επιχειρηματικότητα, η οποία είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, όμως ο σύνδεσμος αυτής ε, με τις αξίες για τις οποίες μιλήσατε είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και υπάρχει μια εύκολη απάντηση σε αυτό, το οποίο είναι να βάλουμε τη λέξη κοινωνική μπροστά από την επιχειρηματικότητα, διότι έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε νέους ανθρώπους οι οποίοι θα δημιουργούν startups, θα, θα επιτυχαίνουν στην επιχειρηματικότητα, όμως ταυτόχρονα θα είναι ενεργοί πολίτες ε, και αξιοπρεπή μέλη της κοινωνίας. Ενώ δεύτερον θα ήθελα να μάθω τις απόψεις σας ε, σχετικά με την καταπολέμηση των φραγμών στην επιχειρηματικότητα ε, και βασικά μαθήματα διότι γνωρίζουμε ότι οι επιστήμονες χρειαζόνται το επιχειρηματικότητα, θα χρειάζονται οραματισμό και να φανταστούν το αδύνατο στο μέλλον και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε αν δεν έχουμε εκπαιδευτεί στις τέχνες για παράδειγμα. Έχει αυτό το λόγο ε, θα ήθελα να επαναφέρουμε τις τέχνες σε αυτό διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ ο Τόμας Μάνιν από την ΙΠΠΗ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θεωρώ ότι είναι σημαντικό το ότι οι δύο επιτροπές μας ε, συνεργαζόμαστε. Όσον αφορά ε, το ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων, είναι το πλαίσιο το οποίο συζητά για τις ικανότητε στην Ευρώπη. Θα θέλαμε λοιπόν ε, αρκετές ικανότητε που υπάρχουν στην Ευρώπη να βγουν από, από το παρασκήνιο. Ε, Ποιε ικανότητε είναι σημαντικέ για την Κομισιόν. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ανταλλαγή απόψεων σε αυτό. Επίσης δεν χρειαζόμαστε και μια ευρω... εξευροποίηση της ε, δυτής εκπαίδευσης που είναι επιτυχημένη σε αρκετά κράτη-μέλη. Πριν από μερικές μέρες ήμασταν στο Silicon Valley, ε, είδαμε την Google και τη Facebook, εκεί η ψηφιακή ε, ικανότητα είναι απαραίτητη, όμως ταυτόχρονα είδαμε ε, και πράγματα τα οποία περιλαμβάνουν και άλλες ικανότητες όπως είναι για παράδειγμα η επιχειρηματικότητα και το να αναλαμβάνει ευθύνε. ευθύνες. Αυτό που μας είπαν στη Google είναι αν είχαμε ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό επίπεδο το οποίο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διδαχθεί. Ε, ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη συνάδελφη. Ευχαριστώ πολύ για το γεγονός ότι ε, υπάρχει επικοινωνία μεταξύ σας, ε, το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω δύο ερωτήματα. Η κυρία Επίτροπος είπε ότι θέλει να βελτιώσει το επίπεδο των ικανοτήτων, ενώ επίσης ανέφερε ότι υπάρχει 20% ικανοτήτων που απουσιάζουν. Έχετε ερώτημα, έχω το ερώτημα αν έχετε ένα χρονοδιάγραμμα για αυτό το ζήτημα. Φέτος έχουμε τα αποτελέσματα της έρευνας του 2015 θα διατεθούν κατά τα τέλη του 2016 και θα δείξουν αν είμαστε επιτυχημένοι στη βελτίωση των ε, ικανοτήτων ιδιωτών όσον αφορά τις γλωσσικές και μαθηματικές ικανότητες. Ενώ θα ήθελα να τονίσω ότι σε όλα τα σχολεία στην Ευρώπη αλλά και στη Τσεχία έχουμε προβλήματα ε, όπου ε, υπάρχουν ε, ε, προβλήματα με μαθητές και θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τους δασκάλους ώστε να μπορούν να εργάζονται ευκολότερα με αυτούς. Από το EPP θα είμαι σε Ένα σχόλιο πριν από 18 χρόνια τελείωσα το σχολείο και θυμάμαι λοιπόν ότι τότε συζητούνταν ότι οι δάσκαλοι θα πρέπει να είναι καλύτερα καταρρισμένοι όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητε και να ρωτιέμαι τι έγινε τα τελευταία 18 χρόνια όταν συνεχίζουμε μιλούμε για αυτό θα ήθελα πιο συγκεκριμένα να πω το ζήτημα της κατάρτασης στην αγορά εργασίας. Η κυρία Τάισεν είπε έναν ε, καλό αριθμό, το 13% των αποφύτων πανεπιστημίου συζητούν, ε, εργάζονται μάλλον σε τομείς που δεν σχετίζονται με αυτό που σπούδασαν ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε σε πάρα πολλούς ε, τομείς, έχουμε υψηλά ποσοστά ανθρώπων που εγκαταλείπουν το σχολείο και αυτό σίγουρα ανέρχεται στα εκατομμύρια, ε, σε δισεκατομμύρια άμα το ε, μεταφράσουμε σε οικονομικούς όρους. Το ερώτημα που έχω λοιπόν είναι πώς μπορεί η Κομισιόν να βοηθήσει ούτω ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν πιο συγκεκριμένα να επικεντρωθούν στην αγορά εργασίας και στις ικανότητες που απαιτούνται. Ευχαριστώ. Και τώρα ο Λουτζι Μάρκενο από το S&D. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις. Προετοιμασία για την απόκτηση των εικονοτήτων στα πλαίσια της επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και απόκτηση γνώσεων από τις πανεπιστημιακές σπουδές ποιο επίπεδο είναι πιο κατάλληλο έτσι ώστε να βοηθηθεί η ε, πρόσβαση του εργαζομένου στην εργασία. Οι μελέτες μέχρι τώρα δείχνουν ότι τα επόμενα δέκα χρόνια θα υπάρξουν δεκάδες νέες επαγγελματικές δραστηριότητες των οποίων η σημασία δεν αναγνωρίζεται από τα συστήματα εκπαίδευσης. Συνεπώς λοιπόν τι κάνετε ως προς αυτό. Και δεύτερη ερώτηση. Μιλάτε για την βελτίωση του πνεύματος της επιχειρηματικότητας. Είπατε ότι θα δαπανίσατε και σημαντικούς πόρους, όπως είπε η Επίτροπος Τάισεν. Εδώ το θέμα της κατάρτισης τίθεται μεν. Από την άλλη όμως υπάρχει και το θέμα των πραγματικών δυνατοτήτων δημιουργίας ε, μιας start-up. Πρόσβαση στην πίστοση υπάρχει. Θα βρίσκουν χρήματα για να ξεκινήσουν. Βρίσκεται λύσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βάντερ Κάντελερε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπατε πολύ σωστά το όνομά μου. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επιμείνει στο πέρασμα από την εκπαίδευση κατάρτιση στην επαγγελματική δραστηριότητα. Είναι σαφές βέβαια ότι οι αρμοδιότητες οι οποίες θα πρέπει να αποκτηθούν <clears throat> θα καλύπτουν και έναν τομέα τον οποίο θα ονόμαζα εγώ ε, μη τυπικό τομέα. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ξεκινήσει δραστηριότητες έτσι ώστε οι νέοι να μπορούν να μεταδίδουν τις αρμοδιότητές τους έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερη θα έλεγα γνώση των ε, ικανοτήτων τους από τους εργοδότες. Η κυρία Τρίπελ. Θα ήθελα να σας θέσω το εξής ερώτημα. Είστε έτοιμοι να αποδεχθείτε ε, τη συμμετοχή οργανώσεων στην ανάπτυξη των ικανοτήτων διότι αυτό απαιτεί ε, το να προσεγγίσουμε νέους ανθρώπους ε, και κυρίως ανθρώπους από, από υποβαθμισμένα περιβάλλοντα και όσον αφορά την εκπαίδευση της επίσημης και ανεπίσημης εκπαίδευσης για την υποστήριξη, των την ανάπτυξη, την υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων για τους νέους και το πώς έτσι θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους από αυτούς οι οποίοι λίγο πολύ ε, είναι σε πλεονεκτική θέση. Ε, e, Τώρα θα ήθελα να μιλήσω τους επιτρόπους. Θα ήθελα να μιλήσω στους επιτρόπους ε, για να τους ευχαριστήσω ε, και χαίρομαι ιδιαίτερω ε, που συνεργάζονται και παρουσιάζουν από κοινού το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η εκπαίδευση λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική και, για την, ε, και στον τομέα της συνεργασίας. Θα, χαίρομαι που αναφερθήκαμε στα σωστά ερωτήματα σήμερα καθώς επίσης και στο ζήτημα της εκπαίδευσης ε, στις ε, βασικές ικανότητες. Κάποιες χώρες στο παράκονον όμως επικεντρώθηκαν ιδιαιτέρως στις ανθρωπιστικές επιστήμες ε, και παραμέλησαν τις θετικές επιστήμες και δεν νομίζω ότι αυτό είναι μια σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει λοιπόν να ανοίξουμε περισσότερο τα εξχολεία μας και το εκπαιδευτικό μας σύστημα σε επιχειρηματικές ικανότητες που θέλουμε να συμπεριλάβουμε και θα πρέπει λοιπόν να διδάξουμε καλύτερες ικανότητες παιδιά μας. Αγαπητοί Επίτροποι, λοιπόν, πιστεύετε ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα έχουν μια καλή επιρροή στα σχολικά μας συστήματα. Και εδώ αναφέρομαι και στην εγγύηση νεολαίας. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους επιτρόπους. Ε, θα ξεκινήσω με την κυρία ε, Τίσν. Πέντε λεπτά όμως. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς σε 5-6 ε, ερωτήσεις ταυτόχρονα μέσως, ε, με, με τόσο λίγο χρόνο. Δεν θα είμαι λοιπόν πάρα πολύ αναλυτική στις απαντήσεις τις οποίες θα σας δώσω. Η ανάγνωση, η γραφή, οι αριθμητικές ικανότητες, αυτές είναι οι βασικές ικανότητες. Τι σκοπεύουμε να κάνουμε σε σχέση με αυτές είναι θα έλεγα αρμοδιότητα αυτών που οργανώνουν τα επίπεδα διδασκαλίας. Τα επίπεδα διδασκαλίας ο λέγει ότι δεν είναι πολύ ικανοποιητικά στην Ευρώπη, δεν είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τα επίπεδα τα οποία χρησιμοποιούμε. Αυτά είναι θέματα βέβαια τα οποία αφορούν στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τις αρμόδιες υπηρεσίες τους. Αυτή είναι υπεύθυνη για την οργάνωση των προγραμμάτων διδασκαλίας. Δεν υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει όμως εμείς στην Ευρώπη να ανταλλάξουμε τις πρακτικές μας <clears throat> να συγκεντρώσουμε όλους τους εμπλεκομένους έτσι ώστε να ωφεληθούν από τις εμπειρίες των άλλων. Και φυσικά απαιτείται να υπάρχει σχέση στενή ανάμεσα στην οικονομική δραστηριότητα από τη μία, τους εργοδότες από τη μία και τα συστήματα εκπαίδευσης από την άλλη. Όταν βλέπει κανείς τα δημόσια συστήματα εκπαίδευσης, όταν υπάρχει ένα κεντρικό όργανο το οποίο ε, επηρεάζει τα, τα προγράμματα διδασκαλίας και στο οποίο συμμετέχουν και εκπρόσωποι και των εργαζομένων και των εργοδοτών, τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Τέτοιου είδους, ε, θα έλεγα, συστήματα βελτιώνουν τις γνώσεις και τις ικανότητες. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα έτσι ώστε οι ικανότητες ατυπικές ή τυπικές των εργαζομένων να είναι ορατές και να μπορούν να τους προσεγγίσουν οι εργοδότες. Εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα κάνουμε ορισμένες προτάσεις έτσι ώστε πράγματι οι ικανότητες να είναι πιο ορατές και πιο αναγνωρίσιμες. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι αναζητούν θέσεις απασχόλησης πέραν των συνόρων μάλιστα, να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και με τις μη τυπικά πιστοποιημένες γνώσεις τους. Εδώ η Ευρώπη έχει κάτι να προσφέρει. Τώρα, για τα συστήματα εκπαίδευσης γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιοι που εγκαταλείπουν τα συστήματα αυτά πρόωρα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ξεκινούν με μειονεκτήματα εξ αρχής και δεν διευκολύνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Εδώ τίθεται το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και οι συστάσεις αναχώρα. Τώρα την κινητικότητα, οι διασυνοριακές σχέσεις, το ότι κάποιες χώρες παρέχουν σωστή εκπαίδευση και εύκολη πρόσβαση στην απασχόληση αυτό είναι κάτι το θετικό που μπορεί να ωφελήσει και τις γειτονικές χώρες. Γιατί, γιατί ζούμε σε μια ανοιχτή αγορά και κάθε κράτος μέλος ωφελείται από τις ικανότητες της ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει όμως παρόλα αυτά το πέρασμα από τη μία χώρα στην άλλη του εργαζομένου να γίνεται με αξιοπρεπή τρόπο. Δεν μπορούμε εμείς ε, να ζητάμε από τους εργαζομένους να είναι κινητικοί και να μην χρησιμοποιούμε και να αμείβουμε σωστά τις ικανότητες που έχουν απεκτήσει σε μια, αποκτήσει σε μια άλλη χώρα. Τώρα για την επαγγελματική κατάρτιση και την τεχνική κατάρτιση λέω στον κύριο Μάννα. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να είναι γνωστές και να κυκλοφορήσουν οι σωστές ε, ε, μέθοδοι ε, δεν υπάρχει επαρκή σεβασμό σε τέτοιου είδους ε, μορφές εκπαίδευσης, την τεχνική εκπαίδευση. Πρέπει λοιπόν να κάνουν προσπάθειες οι Ευρωπαίοι πολίτες περισσότερες από ό,τι σήμερα. Τώρα για τις ικανότητες των διδασκόντων είναι ένα θέμα στο οποίο επανερχόμεθα συνεχώς. Προφανώς οι διδάσκοντες θα πρέπει να έχουν σωστή κατάρτιση. Ε, για τις ψηφιακές γνώσεις. Προφανώς το πρόβλημα υπήρχε πριν 10 χρόνια και υπάρχει και σήμερα. Η πληροφορική έχει, θα έλεγα και η ψηφιακή οικονομία διευρυνθεί τόσο πολύ που τα προβλήματα που έχουμε δεν έχουν καλυφθεί ακόμα πλήρως. Σε επίπεδο λοιπόν αρμοδιοτήτων και ικανοτήτων είναι προφανό ότι θα πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες αυτές και αυτό ισχύει και για τους διδάσκοντες. Μακρηγορώ συνεχώς και ζητώ συνεχώς συγγνώμη γι' αυτό λέει η Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ για την κυρία Ρενά. Έχουμε κάποια πολύ σημαντικά και θεμελιώδη διαγραφή Ευρώπη 2020, τη 2020 τις εκθέσεις επισκόπηση, δήλωση των διακήρυξεων των Παρισίων. Και έτσι προάγονται οι διαστάσει κοινωνική ενσωμάτωσης και για τα εκπαιδευτικά συστήματα. Υπάρχουν λοιπόν πολλές δυνατότητες να τηρηθούν και οι δύο ορίε του Ευρώπη 2020 το 11%, δηλαδή μάλλον το 10% που τώρα εντωμεταξύ έχει φτάσει στο 11%, ο στόχος ήταν 10%. Ωστόσο, για εκείνου που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο το 2020, είμαστε στο 11%, άρα έχουμε τεράστια πρόοδο και θα επιτύχουμε κατά πάσα πιθανότητα το στόχο. Επίσης για την τρίτο βάθμη εκπαίδευση έχουμε στόχους και διορίες και σε αυτά προχωρούμε. Για την Ευρώπη 2020 είμαστε σε αρκετά καλή θέση και μπορούμε να στηρίξουμε τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα στις προσπάθειές τους προς αυτήν την κατεύθυνση. Και η διακήρυξη των Παρισίων και το Ευρώπη 2020, το ΙΤ ε 2020 έχουν στοιχεία και διαστάσεις για κοινωνική ενσωμάτωση και ενίσχυση της πτυχής ενσωμάτωσης μέσα από την εκπαίδευση. Για την κινητικότητα μαθητευομένων. Θα σας υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη έθεσε σε κίνηση ένα πιλωτικό πρόγραμμα του κυρίου Αρτουή. Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για μακροχρόνια μαθητεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο μέσος, όρος, ο μέσος χρόνος μαθητείας με το Erasmus Plus είναι, μάλλον χωρίς το Erasmus Plus είναι δύο-τρεις εβδομάδες, είναι πολύ λίγος. Και τώρα υπάρχει ένα σχετικό πρόγραμμα το οποίο προσπαθεί να εξασφαλίσει και τη συνεργασία των κρατών μελών για πιο μακροχρόνιες περιόδους μαθητείας, από δύο μήνες μέχρι και δώδεκα. Σημαντική βελτίωση λοιπόν. Εάν σε αυτό κατάστημα επιτυχής, θα έχουμε πιστεύω δυνατότητες και από το Erasmus Plus και από το Κοινωνικό Ταμείο πιστεύω να αναπτύξουμε το πρόγραμμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με μακρύτερες περιόδους μαθητείας. Για το STEM και το STEAM συμφωνώ. Πρέπει να καταρριφθούν οι φραγμοί μεταξύ της δημιουργικότητας ε, των πανεπιστημιακών δεξιοτήτων και να ανοίξουν ε, δύο δι μεταξύ των δύο αυτών πλευρών της ζωής. Έχουμε προγράμματα από το Creative Europe, παραδείγματι, έργα του Creative Europe, που μπορούν να αναπτυχθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ε, και Τεχνολογία. με κύριο καθήκον να φέρει σε επαφή το EIT ε, και πανεπιστημιακούς και επιχειρηματίες και ε, φοιτητές ώστε να προωθήσει την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τον επαγγελματικό βίο. Και καθώς η πανεπιστημιακή γνώση πολύ γρήγορα μπορεί να χάσει την επικαιρότητά της, σημασία έχει η ανάπτυξη της διαρκούς επιμορφωσής στις δεξιότητες και κυρίως στις δεξιότητες εκείνες τις κοινωνικές που επιτρέπουν ταχεία προσαρμογή στις ε, ε, νέες κάθε φορά απαιτήσει του επαγγελματικού βίου και σε αυτό ιδιαίτερα υπογραμμίζουμε την σημασία των ε, ικανότητων επικοινωνίας, ε, δημιουργίας ομάδων, όλες αυτές δηλαδή τις κοινωνικές δεξιότητες που θα επιτρέψουν στους νέους να βρουν ένα μια καλύτερη θέση στην κοινωνία, μια πιο σταθερή θέση στην κοινωνία. Συνεργασία με οργανώσεις νέων υποστηρίζω την ιδέα και επιπλέον κάνουμε πολλά. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες ήμουν σε εκδηλώσεις με οργανώσεις νέων. Συγκεκριμένα σε μία συζητήσαμε τα προβλήματα του εξτρεμισμού, της ριζοσπαστικοποίησης, προβλήματα ε, σχετικά με την αγορά εργασίας ε, και την απομόνωση, καθώς πολλές φορές αυτά επικαλύπτονται νέοι που προέρχονται από μειονεκτικό κοινωνικό υπόβαθρο τίνουν περισσότερο προς την ριζοσπαστικοποίηση και τις πολιτικές ε, εξτρεμιστικές δυνάμεις αφενός, αφετέρου δε. Δυσκολεύονται να βρουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Δεξιότητες λοιπόν, κατάλληλες δεξιότητες, αποτελεσματική εκπαίδευση, και εξασφάλιση για τους νέους των κατάλληλων δεξιοτήτων. Αυτά είναι τα καλύτερα εργαλεία για την πολιτική και κοινωνική σταθερότητα και βέβαια οι οργανώσεις των νέων είναι παράγον σοβαρός στην προσπάθεια αυτή. Και βεβαίως υποστηρίζουμε πολλά προγράμματα γεφύρωσης μεταξύ της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Έχουμε προγράμματα βάσης μέσα στο Erasmus Plus, παραδείγματι. Έχουμε χαρτογράφηση για το κοινωνική ενσωμάτωση, κοινωνικό αποκλεισμό με την υποστήριξη σε θέματα πολιτισμού. Και ενθαρρύνουμε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να ανοίξουν τις δομές τους. και σε πιο και σε λιγότερο τυπικές ή και άτυπες μορφές εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ τους Επιτρόπους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω, γιατί δεν έχουμε πια χρόνο, δύο τελικές παρατηρήσεις. Ξεκινώντας, να πω ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να υπάρξει μια μέθοδος εργασίας η οποία να συμφωνηθεί και με τους συναδέλφους της άλλης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής μια πιο εγκάρσια αν θέλετε και ε, σφαιρική αντιμετώπιση αυτού του πακέτου. Ε, γιατί έχουμε και οι δύο επιτροπές αρμοδιότητα εδώ. Πρέπει να συνεργαστούμε λοιπόν. Αυτό γίνεται και σε επίπεδο ε, Συμβουλίου Υπουργών, όπου γίνονται συστηματικές συναντήσεις και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της συνεργασίας των δύο επιτρόπων και γενικών διευθύνσεων. Έτσι θα διασφαλίσουμε τη συνέχεια που απαιτείται δεύτερον. Και έγινε μια κάποια αναφορά χωρίς όμως να υπάρξουν πάρα πολλές διευκρινήσεις. Τι διαβουλεύσεις γίνονται στην παρούσα φάση. Είναι διαβουλεύσεις των κοινωνικών εταίρων, συμμετέχουν οι οργανώσεις των νέων, συμμετέχουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και μία τρίτη ερώτηση, παρατήρηση. Παρουσιάστηκαν προτάσεις, ακροάσεις για την διοική λεγόμενη κατάρτιση εκπαίδευση και για την πρόσβαση στην κατάρτιση. Θα πρέπει εδώ, όπως έλεγαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, να είναι μέτρα ενσωματωμένα στο σύνολο ευρύτερων πολιτικών, κατά πολέμηση της φτώχειας, κάλυψη των μειονεκτικών ομάδων και ιδιαίτερα των ομάδων των πολιτών με αναπηρία κτλ. Εδώ τα εκπαιδευτικά συστήματα μέλη να κάνουν πολλά. Η επικουρικότητα υπάρχει, αλλά τι σημαίνει. Σημαίνει μεν σεβασμός των αποφάσεων των εθνικών συστημάτων παιδείας, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το ανοιχτό επίπεδο, η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού και στα πλαίσια των στόχων της στρατηγικής 2020 και μέσω των συστάσεων του εξαμήνου που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε τα μέτρα μας ε, να είναι πιο αποτελεσματικά και να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός χώρος καινοτομίας στην απασχόληση ίσων ευκαιριών για όλους. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Πάνω σε αυτό λοιπόν και έχει σημασία να δούμε τι δεδομένα έχουμε στην διάθεσή μας, μία από τις προτάσεις μας είναι η αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας με ποιο τρόπο θα γίνει θα το δούμε. Και δεύτερον η εκπαίδευση έχει διπλή φύση. Από τη μία προετοιμάζει τις γνώσεις των πολιτών αλλά και την απασχολησιμότητά τους. Οπότε τα συστήματα μεταξύ τους θα πρέπει να επικοινωνούν καλύτερα. Το πρόβλημα είναι ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα dual education, διοικής κατάρτισης, εκπαίδευσης. Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά συστήματα με διαφορετική αποτελεσματικότητα. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα γιατί η φτώχεια στην κατάρτιση και η έλλειψη βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων οδηγούν στην φτώχεια και στην ανεργία. Δεν αρκεί βέβαια η επαγγελματική κατάρτιση, αν δεν υπάρχει και μια δυνατότητα διεύρυνσης των βασικών γνώσεων και ικανοτήτων των πολιτών. Γιατί η ταχύτατη αλλαγή των αγορών εργασίας τελικά δεν επιτρέπει στους εργαζομένους να προσαρμοστούν και να προβλέψουν εκ των προτέρων τις εξελίξεις στην απασχόλησή τους. Εδώ η διαβίου κατάρτιση δίνει λύσεις. Ε, τα μέσα λοιπόν που έχουμε στη διάθεσή μας είναι γνωστά. Αναφερθήκατε σε αυτά εσείς στην πρώτη σας παρέμβαση, η Επίτροπη εννοώ. Πρέπει όμως να είμαστε λίγο πιο δημιουργικοί και λίγο πιο θαραλέοι. Η συμμαχία για την γνώση, οι εταιρικέ σχέσεις ανάμεσα στην κατάρτιση, την εκπαίδευση, την έρευνα, και την οικονομία. Και από την άλλη έχουμε προγράμματα όπως το Erasmus Plus που επιτρέπει να γίνουν θετικά βήματα. Η αναγνώριση των μη τυπικών, των ατυπικών γνώσεων δεν είναι κάτι το οποίο έχει ολοκληρωθεί από πλευράς μας. Ως εκ τούτου λοιπόν, χωρίς αυτές τις κομβικές ικανότητες, χωρίς τη δραστηριοποίηση του ίδιου του πολίτη, δεν μπορούμε να έχουμε την απαιτούμενη επιθυμητή απασχολησιμότητα. Και τίθεται τελικά και το θέμα των οικονομικών πόρων. Χωρίς αυτό δεν υπάρχουν τα άλλα. Τα διάφορα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα μέσα που τους δίδει η πολιτική συνοχής, πρέπει να υπάρχει σωστός διαμερισμός των στρατηγικών αλλά πρέπει να γίνει και σωστή χρήση του στρατηγικού επενδυτικού ταμείου. Είναι, θα έλεγα, το αποτέλεσμα μέχρι τώρα της παρέμβασης του στρατηγικού αυτού ταμείου, του Juncker Plan, όπως λέμε, ανεπαρκές. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να στηρίξουμε τα μέτρα μας με πιο συγκεκριμένο τρόπο γιατί αλλιώς θα παραμείνουμε θεωρητικοί και μόνο. Ευχαριστώ λοιπόν τους δύο επιτρόπους και εξ ονόματος της συναδέλφου Προέδρου και ελπίζω να γίνουν και άλλες τέτοιου είδους πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις. Ευχαριστώ φυσικά και την επιμελητία, διερμηνής, γραμματεία κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης ότι έχουμε άλλα δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη για σήμερα. Γι' αυτό το λόγο θα σας παρακαλούσα να παραμείνετε αφορά ε, το Κοινωνικό Ταμείο καθώς επίσης ε, και το Ταμείο Προσαρμογής θα ήθελα τους συντονιστές ε, της Επιτροπής Πολιτισμού να πάνε στην αίθουσα 3G2.